Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω, να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Θέλω να είμαι ακριβής, λίγο πολύ. Σημείο ένα τη διάταξης είναι η έγκρισή της. Μήπως έχετε αντιρρήσεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Δεν νομίζω. Εν τη αυτή περιπτώσει εγκρίνεται η μυρίσια διάταξη ως έχει. Ορχόμαστε λοιπόν στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης που αφορά τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Καταρχάς, καλωσορίζω τέσσερα νέα μέλη που καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Δεν βλέπω τον συνάδελφο, τον κύριο Νεγκρέσκου από τη Ρουμανία και τον Μάρκο Ζέμπελ από την Ισπανία, σοσιαλιστών. θα έρθουν το πρωί και τον κύριο Μαρίες Μπότος από το Ρινιού, από τη Ρουμάνια. Και Αλάνα Σικαρέλ από τη Γαλλία, από το Ρινιού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και είσαστε μέλη της ομάδας μας, της Επιτροπής μας. Για διαρμηνία έχουμε τις εξή γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, ουγγρικά, λετονικά, πολωνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και κροατικά. Να σας πω ότι θα έχουμε και αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου της συνεδρίασής μας. Πάμε τώρα στις αποφάσεις ε, των συντονιστών ε, της 21ης Ιανουαρίου του 2021. Σύμφωνα με τις ε, αποφάσεις των συντονιστών, Έστειλα ένα email σε όλα τα μέλη της ομάδας μας, της Επιτροπής μας και στις 24 Ιανουαρίου θα έχουμε την ε, προθεσμία για τις ε, για το θέμα αυτό. Να σας ε, μιλήσω τώρα για το ε, θέμα, ε, το πρώτο της μερισσής διάταξης που έχει να κάνει με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρ Μισελ, έχει προτείνει μία γραμμή συμβιβασμού. Ε, όμως εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη, είναι no-go αυτό που προτείνεται από την πλευρά του Συμβουλίου. Για το Erasmus Plus ε, ε, ε, υπάρχει μια πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρξει τριπλασιασμός των κονδυλίων, το ίδιο και από την πλευρά της Κομισιόν. Αναφέρεται ανάγκη για δραματική αύξηση των κονδυλίων, γιατί και τα πανεπιστήμια και τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα χρειάζεται αυτά τα χρήματα. Εχθές με το συντάκτη της έκθεσης είχαμε μια συνέντευξη τύπου όπου αναφέρθηκε ακριβώς αυτό το θέμα ε, και είπαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικά με το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν χαιρετίζουμε τις τρεις ε, πρωτοβουλίες που έχουν έρθει από την πλευρά του Κοινοβουλίου, όμως χωρίς τα απαραίτητα χρήματα είναι τρελό, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν καλά προγράμματα ε, τα οποία λειτουργούν καλά και στο Συμβούλιο και τα οποία ε, δεν έχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Εμείς ε, δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά την Κυριακή και τη Δευτέρα να τα ξεχνάμε ως πολιτικοί. Είναι σημαντικό να λέμε πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η ανταλλαγή φοιτητών, οι πολιτιστικές ανταλλαγές. Αυτά είναι σημεία που μας βοηθούν να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια, τα χρηματοδοτικά μέσα, ένα... Ε, έχουμε φυσικά επενδυτικά ταμεία, έχουμε τη γεωργία, έχουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά χρειαζόμαστε και γι' αυτό το θέμα χρήματα. Ως Επιτροπή, λοιπόν, πολιτισμού. Δεν μπορούμε αυτό να το δεχτούμε. Παρακαλώ κινητοποιηθείτε, βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους, να έχουμε όποια υποστήριξη μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο και κοιτάξτε και προς την Κομισιόν. Ούτε η Κομισιόν είναι ικανοποιημένη με αυτά που προτείνεται. Τόσες καλές πρωτοβουλίες που είχε προτείνει η Κομισιόν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτόν τον προϋπολογισμό τα προγράμματα εκπαίδευσης αλλά και το Greater Europe. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Για το Greater Europe δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ε, νούμερα, όμως υπάρχουν κάποιες περικοπές που φαίνονται μέσα στην πρόταση προϋπολογισμού. Και νομίζω ότι έτσι όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, με την κατανομή που έγινε, θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν ε, στην περίπτωση αυτή, ε, όπως και στην περίπτωση του Εράσμους, ε, δεν είναι εύκολο να έχουμε να γίνει τίποτα αν δεν έχουμε την υποστήριξη σε επίπεδο κονδυλίων. Υπάρχει μαζική υποχρηματοδότηση σε κάθε είδους σχέδιο που υπάρχει για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Υπάρχει μεγάλη πίεση λοιπόν προς τα προγράμματα και φυσικά δεν μπορούν να ληφθούν πρωτοβουλίες, ούτε καν να το σκεφτούμε όταν δεν έχουμε χρήματα ε, για να επεκτείνουμε τέτοια προγράμματα και να τα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιο αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίση ως προς την εκπαίδευση και τον πολιτισμό ε, και φαίνεται ότι δεν έχουμε μάθει τα μαθήματά μας. Ε, αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι για το πρόγραμμα Greater Europe είμαστε πιο κάτω από ό,τι ήμασταν. Είναι πραγματική περίπκοπη. Και φυσικά ε, αυτό συνοδεύεται από τη μαζική υποχρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι η δική σας υποστήριξη και συνεργασία είναι απαραίτητη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ε, προχωρήσουμε σε κάποιες προτεραιότητες, να διορθώσει ο Σαλμισελ αυτά που έχει προτείνει και φυσικά να κοιτάξουμε και για την υποστήριξη της Κομισιόν, γιατί έτσι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Äh Συγγνώμη που θυμώνω, αλλά καταλαβαίνετε ε, υπάρχει και το θέμα των χρημάτων και για την έρευνα ε, και τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι και λέμε ότι θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι στην έρευνα και στην ανάπτυξη και μετά κόβουμε τα κονδύλια. Πραγματικά το είπα και χθε. Αν δεν είμαστε υπεύθυνοι άμεσα για την ε, έρευνα, πραγματικά θα έχουν πρόβλημα τα πανεπιστήμια και γενικά δεν θα μπορέσουμε να ησυχάσουμε σε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Έχουμε λοιπόν σήμερα τις ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020. Ήμουνα η εισηγήτρια και γι' αυτό θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Σε αυτό το σημείο να πω στους συντονιστές και τα άλλα μέλη ότι τους ευχαριστώ θερμά για την επικοδομητική συνεργασία. Είμαι πολύ ε, πεπισμένη ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και επειδή έχουμε απτές προτάσεις στο τραπέζι και αν δεν θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι μπορώ να πάμε, μπορούμε να πάμε άμεσα στην ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί. Βάλτε ε, στην υποδοχή. Παρακαλώ. Ξεκινάμε. Παράγραφος 1. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ich schließe die Abstimmung. απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Φαίνεται ότι πάλι την ίδια πλειοψηφία έχουμε, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στη συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά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 να το ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Γιατί είναι ισοψηφία. Πάμε στην τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47. Δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Πάμε στην 48. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα. Ονομαστική ψηφοφορία τελική ψηφοφορία για, τη συνολική, για το συνολικό σχέδιο γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Με μία ψήφο κατά και 23 υπέρ, δύο αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Φτάνουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα Έχουμε εξέταση του σχεδίου γνωμοδότηση για τι κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό του 2021. Τον Δεκέμβρη η Επιτροπή Προπολογισμού αποφάσισε ότι ε, θα αλλάξει το σχέδιο του εσωτερικού προπολογισμού. Έτσι λοιπόν ε, η επιτροπές όπως η Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να εκφραστούν για τα συγκεκριμένα θέματα που τις αφορούν για να, μπορούν, ε, να, μπορεί να θεσπιστεί η διαδικασία προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο. Παρακαλώ σας ζητώ να ησυχάσετε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Κίντο. Με αυτή την ε, απόφαση θα είναι πιο αποτελεσματική η πολιτική που έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές τους. Για το ε, σχέδιο προϋπολογισμού 2021 έχουμε μία γνωμοδότηση με συντάκτη τον Ρωμαίο Φραντς. Έχουμε λοιπόν 21 ε, Φεβρουαρίου την, ε, στις 12 η ώρα την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα έχουμε μια πολύ σύντομη διαδικασία. Ε, αυτό πρέπει ε, να το ξέρετε. Δίνω το λόγο στον Ρωμαίο Φράντς ως ε, εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα για την να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης που έχω ετοιμάσει για την Επιτροπή Πολιτισμού ε, και χαίρομαι και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ε, στο υπόβαθρο αυτής της ε, πρότασης υπάρχει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν κάποια κονδύλια που προβλέπονται συγκεκριμένα για την ε, πολιτισμό και υπάρχουν συγκεκριμένες περικοπές. Θεωρώ ότι είναι εντελώς απαράδεκτες η σημασία των προγραμμάτων στον τομέα της ε, εκπαίδευσης και του πολιτισμού πρέπει ε, να πάνουν μεγαλύτερη έμφαση. Θα έπρεπε να υπάρχει αύξηση τα προγράμματα εκπαίδευσης και πολιτισμού προσφέρουν πολλά σε επίπεδο ε, ακόμα και της, στο επίπεδο ακόμα και της κλιματικής αλλαγής. Όπως γνωρίζετε, οι χρηματοδοτικές ε, ε, τα χρηματοδοτικά μέσα για το Erasmus Plus έχουν μειωθεί σημαντικά και εμείς έχουμε προτείνει σημαντική αύξηση και αυτή συνίσταται σε τρίπλασιασμό των κονδυλίων. Επίσης, ε, αυτά που βλέπουμε σε επίπεδο 2021 είναι σε σχέση με το 2020 όχι μόνο ε, υψηλότερα τα ποσά, αλλά ε, έτσι διαρθρωμένα ώστε να έχουμε καλύτερη επίπτωση. Αυτά τα προγράμματα ε, μεταξύ άλλων και αυτό που υποστηρίζει τον οπτικοακουστικό τομέα, τον ε, ε, δημιουργικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν διπλασιασμό των κονδυλίων τους. Υπάρχουν κάποια σχετικά νέα προγράμματα, αυτά για την ελληνική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά βλέπουμε ότι σε σχέση με, το, με την πρόταση της Κομισιόν είναι ίδια τα ποσά. Επίσης, Έχουμε πολλές προσδοκίες ε, σχετικά ε, με αυτά τα προγράμματα, ειδικά για τους νέους στην Ευρώπη. Έχουν μεγάλες προσδοκίες από το πρόγραμμα. Επίσης, η εμπλοκή των πολιτών ε, στα προγράμματα αυτά θα πρέπει να συνοδεύεται από μια χρηματοδοτική υποστήριξη ε, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ισότητα, ε, τη συμμετοχή των πολιτών ε, στις αξίες της Ευρώπης. Υπάρχουν έξι σημεία στις τροπολογίες μου, τα οποία θα ήθελα τώρα να θίξω. Καταρχάς, άλλη μια φορά, τονίζω τη σημασία των προγραμμάτων για τους κοινωνικούς στόχους, ειδικά για την συμπερίληψη όλων των ανθρώπων. Το τονίζω αυτό. Επίσης, ε, ο ρόλος των προγραμμάτων ε, στην ε, κλιματική αλλαγή, στην αλλαγή νοοτροπία στο περιβάλλον είναι πολύ σημαντικός. Φαίνεται μέσα από τις τροπολογίες μου. Για τα πιλωτικά προγράμματα ζητώ από την Κομισιόν να υπάρχει ε, έγκαιρη κατάθεση του ε, χρονικού πλαισίου με διαφάνεια. Επίσης, για προγράμματα όπως το EFSE και τον Ορίζοντα 2020, ζητώ από την Κομισιόν να έχει πιο συνεκτικές στρατηγικές, έτσι ώστε τα προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της, ε, των δημιουργικών τεχνών να είναι πιο αποτελεσματικά. Να ήθελα επίσης να πω ότι αν είχαμε, αν είχαμε επανάληψη του πολιτούς δημο, δημοσιονομικού πλαισίου που λύγει τώρα, ε, δεν θα είχαμε τα σωστά αποτελέσματα. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις ε, που ε, άτομα και μικρές επιχειρήσεις, μικροί οργανισμοί μάλλον, στηρίζονται σε αυτά τα κονδύλια και δεν πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ των δύο πλαισίων. Τέλος, πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη επικοινωνία ε, για όλα τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποστηρίζουμε μια τέτοια προσέγγιση. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι για την υποστήριξη της γνωμοδότησής μου και θα δεχτώ με χαρά τις τροπολογίες σας. Ευχαριστούμε, Φραντς. Ξεκινάμε με το σκιώδη συγητή, τους σκιώδης εισηγητές. Εσύ μιλάς εκ μέρους του Έλερ. Η κυρία Φεράντη είναι πρώτη, μετά Σλαμπάκοφ, Έλερ, Πετραβέρ. Μιλάει για σας. Ποιος μιλάει για σας. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Ωραία. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να υποστηρίξω την πρότασή σας, την αρχική όσον αφορά το προπολογισμό για το ΣΥΝ είναι πραγματική πηγή κινητοποίησης. Θέλω να επαναλάβω ότι συμμερίζομαι αυτά που είπατε όλα. Είμαστε στη διάθεσή σας για να δώσουμε αυτή τη μάχη που είναι πρωταρχική σημασία όσον αφορά τους στόχους μας για την παιδεία και τον πολιτισμό. Να ευχαριστήσω τον Ρωμαίο Φραντς. Πολύ καλή δουλειά έκανε ως εισηγητής. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες είναι όλες χρήσιμες και σκόπιμες και θα ολοκληρώσουν το σχέδιο γνωμοδοτήσεως διατηρώντα το κείμενο βραχή, υπενθυμεί τι προτεραιότητέ μα στον προπολογισμό, υπογραμμίζονται σημαντικέ πτυχέ, όπω η ανάγκη που προσαρμόσουμε τα προγράμματα στην αργή τη κοινωνία και την πρόκληση του περιβάλλοντο. Υπογραμμίζει και κάποιε πτυχέ πιο πρακτικέ, όπω είναι σημασία να, πληρών, να γίνονται πληρωμένε συμμετέχοντε και να αξιολογούνται ταχύτερα οι προπαρασκευαστικέ δράσει και τα πιλωτικά προγράμματα. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα υποστηρίξουμε αυτή την γνωμοδότηση και κάποιες τροπολογίες που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε θα ενταχθούν με σωστό τρόπο στο σχέδιο κειμένου. Ευχαριστώ. Äh, äh, Ευχαριστούμε τη Λοράνς Φεράν. Κύριος Λαπάκοφ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ίσως σας εκπλήξει αυτό που θα πω ανήκω στο ECR, αλλά θα πω ότι είναι πολύ καλή έκθεση. Δεν θα αναφέρω όλα τα στοιχεία τα θετικά που μου αρέσουν. Είναι αρκετά εξαντλητικό το κείμενο, περιέχει πολλά. Η παρουσίαση ήταν διεξοδική που έκανε ο συνάδελφος. Να μιλάω πιο σιγά. Εντάξει. Συγγνώμη. Εν κατακλείδη, μου αρέσει πολύ η έκθεση και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που έχουμε παρόμοια προσέγγιση. Σκεφτόμαστε ε, παρόμοια πράγματα. Αυτό που πρέπει να διορθωθεί κατά την άποψή μου είναι ότι πρέπει να τριπλασιαστεί ο προπολογισμό για την Ευρώπη, όχι να διπλασιαστεί. Το μόνο πρόβλημα είναι τα προγράμματα για τον πολιτισμό, την παιδεία και τη δημιουργικότητα και πώς μέσω των προγραμμάτων θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της αλλαγής του κλίματος. Ίσως χρειάζεται καλύτερη διατύπωση το κείμενο. Εκεί. Πρέπει να τονίσουμε περισσότερο το ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα είναι φορείς οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Σχετίζεται με τους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει η κοινωνία μας. Και όταν ένα πρόγραμμα είναι τόσο επιτυχές όπως το Erasmus ΣΥΝ, πρέπει να διευρύνεται και όχι να συρρυκνούται όπως προτείνεται. Ή να τίνει να εξαλειφθεί λόγω ελλείψους χρηματοδότησης. Πρέπει να έχουμε περισσότερους πόρους. Σημαντική αύξηση χρειαζόμαστε. Ίσως πρέπει να συντάξουμε μια επιστολή ή να βγούμε στους δρόμους να το διαλαλήσουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε χρήματα για τον πολιτισμό και για την παιδεία. Και είναι ένα μάρτυμα που κάναμε όλοι οι πολιτικοί, σε όλες τις χώρες. Τα πρώτα χρήματα που αφαιρούν είναι για τον πολιτισμό και την παιδεία. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Ευχαριστώ. Μιχαήλα Γιώργοβα. Είναι η εκπρόσωπο του κυρίου Έλλερ. Ε, Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Λέερ στηρίζει την α, γνωμοδότηση. Να στηρίξω κάτι, να υποστηρίξω κάτι. Πιστεύω ότι οι προσεγγίσεις μας συμφωνούν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα στείλω επιστολή στον κύριο Μπάμπιτς, τον πρωθυπουργό μας, και θα του ζητήσω στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να απορρίψει την πρόταση του Προέδρου α, του Συμβουλίου του κ. Σαλμισελ που προτείνει σημαντική μείωση των πόρων για το έρασμος και επίση μείωση των στόχων στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας. Είναι μια δραστηριότητα που ενδιαφέρει και θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτό ο Πρωθυπουργό μας. Ίσως έχετε άλλες ιδέες. Η πρόταση που κάνει ο συνάδελφος ε, οι προτάσεις που κάνει με βρίσκουν σύμφωνοι, τις υποστηρίζω και όσον αφορά το έρασμος, αυτό αφορά επένδυση στη νέα γενιά. Είναι ένα πρόγραμμα συμπεριληπτικό και θα θέλουμε να μην είναι αποκλειστικό και να εξαιρούνται άνθρωποι από το Εράσμος. Να μην απορρίπτεται σημαντικό ποσοστό των προγραμμάτων, να είναι συμπεριληπτικό πρόγραμμα, κυρίως για τους νέους, τους νέους που δεν έχουν τη δυνατότητα, τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχουν δεν έχουν τη σωστή πλαισίωση. Αυτό σχετίζεται με τη δημιουργικότητα, με αξίε όπως είναι η αλληλεγγύη. Γι' αυτό η πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου για μας δεν μπορεί να υποστηριχθεί και η θέση του συναδέλφου εν ονόμα της Επιτροπής μας είναι κάτι που θα υποστηρίξω πλήρως. Η κυρία Πέτρα Κάμερ Εβερτς, ε, εκπρόσωπος ε, του κυρίου Νεμπρέσκου, ε, του κυρίου ε, ο κύριος Νεκρέσκο ζητά συγγνώμη. Έπρεπε να επιστρέψει στη χώρα του. Μα δώσω λοιπόν την εντολή των εκπροσωπήσω. Χαιρετίζουμε τη γνωμοδότηση του εισηγητή. Ε, όλα τα σημαντικά σημεία για μας αναφέρονται στη γνωμοδότηση και ε, Επίσης ε, το υπόβαθρο ε, το οποίο παρουσίασε η Πρόεδρος ε, είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνους. Θέλουμε φυσικά να εμποδίσουμε στην αρχή του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2001-2027 να υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή των κονδυλίων. Ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε σε αυτό το σημείο να ζητήσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να ξεκινήσει όντως τον Ιανουάριο το πρόγραμμα και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα θα λειτουργήσουν ομαλά. Και ελπίζουμε ότι μέχρι τον Νοέμβρη ε, θα έχουμε καταφέρει να αποφασίσουμε τα σχετικά εδώ σε αυτό το σώμα για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιο διάστημα, ένα μήνα και, ε, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά ε, όλες οι προετοιμασίες ε, και να δίνονται τα χρήματα και για το Erasmus Plus και για το Creative Europe και για το πρόγραμμα για την ελληνική στην Ευρώπη και να ξεκινήσουν όλα ακριβώς το Γενάρη του 2021. Επίσης, ε, για τα μέτρα που αφορούν ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και την επικοινωνία, θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να είναι στο μέλλον λίγο διαφορετική η στάση της από ότι στο παρελθόν. Υποστηρίζουμε λοιπόν τον συνάδελφο σε όλα όσα έχει προτείνει και θα θέλαμε να τονίσουμε λίγο ένα-δύο σημεία, ειδικά το θέμα των του σχεδίου έκτακτης ανάγκησης έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να πετύχουμε τους κοινωνικούς στόχους της Ευρώπης και τα προγράμματα ε, να μην είναι απλώς εκεί για το φαίνεστε, αλλά να έχουν τη συμβολή που πρέπει για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να λάβουν το λόγο, η κυρία Σεκουρέλη. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι που Παρίσταμε στην Επιτροπή σας, λυπούμε που συμβαίνει αυτό σε αυτό το πλαίσιο. Μπορείτε όμως να βασιστείτε στην αγωνιστικότητά μου. Είμαι στοχοπροσιλωμένη. Δεσμεύομαι να, να δουλέψω να πετύχω όλους τους στόχους σας. Ε, προσυπογράφω κάθε λέξη που είπαν τα χείλη σας. Και να ξέρετε ότι τις τελευταίες μέρες έχω έρθει σε επικοινωνία με τη γαλλική πλευρά ε, σε σχέση με τον προπολογισμό, ο οποίος υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με τις προσδοκίες μας. Θα υπάρξει κινητοποίηση και θα υπάρξει επίδειξη αλληλεγγύης από την πλευρά του γαλλικού κράτους, των, των επίσημων γαλλικών αρχών, οι οποίες θα κινητοποιηθούν για να σταθούν πλάι μας στις διεκδικήσεις μας. Ευχαριστώ. Μίλαν Σφέρ. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή για όλα όσα είπε σχετικά με το Erasmus Plus. Ε, θεωρώ ε, λοιπόν ότι είμαι υποχρεωμένος ε, να πω κάποια λόγια για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την γνωμοδότηση και για την, την οποία πλήρως υποστηρίζω. Είμαστε όλοι υπέρ μιας αύξησης ε, των ε, χρηματοδοτικών μέσων και φυσικά των κονδυλίων και φυσικά η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι το Erasmus Plus είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Μετά όμως από, τις την εκλογή της έβγαλε άλλο χαρτί και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θέλουμε περισσότερη ε, συμπερίληψη και την εκτέλεση όλων των μεγάλων πρωτοβουλειών που έχουν προταθεί. Ε, έτσι λοιπόν, συμφωνώ πλήρως με όλους τους συναδέλφους ε, και θεωρώ ότι πρέπει να απαιτήσουμε πολύ περισσότερα ε, κονδύλια από όσα έχει προτείνει ο Σαρλ Μισελ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο που να θέλει το λόγο. Δίνω λοιπόν τώρα ε, το μικρόφωνο στην Κομισιόν για να μπορέσει να μας ε, καταθέσει και αυτή τις απόψεις της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τα λεγόμενά σας και προσδίδει τεράστια σημασία στη γνωμοδότηση αυτής της Επιτροπής σε ό,τι έχει να κάνει την νεότητα, την νεολαία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κουλτούρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να σας ε, απευθύνει ένα θερμό ευχαριστώ για την αταλάντευτη στήριξή σας στο πρόγραμμά μας σε αυτούς τους τομείς και σας ευχαριστεί για την έκκληση που απευθύνεται να ενισχυθεί ο προεπιολογισμός για το Erasmus Plus και για τη Δημιουργική Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να αφιερώσουμε ακόμα περισσότερα κονδύλια από ό,τι έγινε αυτό στο παρελθόν και ειδικότερα από το 2014 και μετά, έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά στο μέλλον να μπορέσουν να πετύχουν γρήγορα τους στόχους που επιδιώκουν για περισσότερη κοινωνική συμπερίληψη, για περισσότερους συμμετέχοντα συμμετέχοντες για μεγαλύτερη στήριξη των ατόμων από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με σκοπό ο χώρος της εκπαίδευσης να καταστεί μια απτή πραγματικότητα για την νεολαία μέχρι το 2025, με σκοπό να αναπτυχθούν πλήρως οι πανεπιστημιακές πρωτοβουλίες στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης απανταχού στην Ευρώπη, σφυριλατώντας ισχυρές συμμαχίες, θέλοντας επίσης να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, όπου και αν βρίσκονται και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε στη ζωτικότητα και στην ανάπτυξη και στην άνθηση ε, αυτού του τεράστιου οικονομικού κλάδου που είναι η βιομηχανία του θεάματος, της κουλτούρας, του πολιτισμού και των έργων Με αυτό το πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2018 είχε καταρτήσει μια πολύ εμπεριστατωμένη πρόταση, πολύ προσεκτικά μελετημένη στο πλαίσιο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος, προβλέποντας σημαντικές αυξήσεις στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων μας. Φτάνουμε τώρα σε ένα λεπτό σημείο στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. δε μου μένει παρά να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό αυτή την έκκληση που απευθύνεται για τις περικοπές που ε, επιθυμούν κάποιοι ε, στις πολιτικές μας που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Επίσης, ο χρόνος πιέζει. Και πάνω από όλα αυτό το οποίο ελπίζουμε είναι να επιτευχθεί συμφωνία και εντός Συμβουλίου αλλά και μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το σύνολο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό είναι ζωτική σημασία προκειμένου τα 37 προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να λειτουργήσουν μελλοντικά και να είναι πλήρω λειτουργικά δηλαδή από την 1η του επομένου Ιανουαρίου. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εφαρμογή του υφιστάμενου πολιετούς δημοσιονομικού δημοσιονομικού πλαισίου είχε ήδη, και το επιθυμήσατε κι εσείς, υποστεί σημαντικές καθυστερήσεις οι οποίες αποδείχθηκαν αρκετά επισφαλείς, αρκετά επιζήμιες για πολλούς δικαιούχους των προγραμμάτων μας και για δικαιούχους του Erasmus Plus και δικαιούχους της ε, Δημιουργικής Ευρώπης αυτή, αυτός ο κίνδυνος δεν είναι εικονικός, είναι αληθινός. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να ξεπεράσουμε ακόμα και τις καθυστερήσεις που γνωρίσαμε όταν ε, ξεκίνησε το υφιστάμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να εφαρμόζεται. Μια τέτοια καθυστέρηση και η αμφισημία και η βεβαιότητα και το κατά πόσο θα υπάρξουν και πώς θα εφαρμοστούν τα προγράμματα είναι πάρα πολύ επιζήμια και ε, θα οδηγήσει σε πάρα πολλούς συμμετέχοντες να αποχωρήσουν, ειδικότερα αυτούς οι οποίοι προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε ό,τι ε, αφορά στο προφίλ του προγράμματος Erasmus Plus και τις πιστώσεις πληρωμών σημειώνουμε πολύ προσεκτικά το αίτημα της δικής σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σημειώνουμε επίσης το μέλημά σας. Εσείς θέλετε να διασφαλίσετε μια πρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των δύο ε, περιόδων προγραμματισμού. Να περάσουμε από τη μία στην άλλη απρόσκοπτα. Και το χρηματοοικονομικό προφίλ του κάθε προγράμματος εξαρτάται απολύτως από την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Αυτό πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς ε, για το γεγονός ότι ε, ε συμμερίζεστε την απόψή μας ε, για τον προπολογισμό, ότι υπάρχει ανάγκη για αύξηση, γιατί όλα αυτά τα μέσα είναι σημαντικά για την... Ε, καθυστέρηση στο πρόγραμμα, ο προπολογισμό είναι το ένα κομμάτι. Ελπίζω η Κομισιόν λοιπόν ε, να κάτσει γρήγορα ε, στο τραπέζι με το Κοινοβούλιο για να βρεθεί μια λύση για το θέμα της διακυβέρνησης. Ε, νομίζω ότι η επίτροποι πρέπει να ε, είναι και αυτοί ε, σε συνένεση μεταξύ τους για διάφορα τέτοια θέματα και για τις διαδικασίες ε, και εμείς ως συνομοθέτες πρέπει να επιμένουμε. Κάποιες φορές δεν μπορούμε δηλαδή να παρετούμαστε από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρώπης καθώς εμείς είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι τους και έχουμε την υποχρέωση έναντι των εκλογέων μας να είμαστε πιστοί στις Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κάνουμε μικρή, ένα μικρό διάλειμμα να έρθουν οι εκπρόσωποι που θα προσιάσουν το επόμενο θέμα. Ναι, κάνουμε μια σύντομη διακοπή μέχρι να έρθουν οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος Αναλίντ. Και θα τελειώσουμε πιο γρήγορα φαίνεται. Αλλά να ξεκινούσαμε και λίγο πιο νωρίς. Σταματάμε μέχρι παρατέταρτο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς, για να έχουμε και λίγο χρόνο για την επιτροπή. Λοιπόν, αξιότιμοι συνάδελφοι, σας ζητώ να λάβετε τις θέσεις σας. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, γιατί υπήρξε μια τεράστια ουρά κάτω στην είσοδο από επισκέπτες που έπρεπε να μπουν και ήταν δύσκολο να εισέλθει κανείς γρήγορα στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, ε, με χαρά μου καλωσορίζω τους ε, εκπροσώπους ε, από το Ίδρυμα Αναλύτ. Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα Erasmus for Associations ε, ε, το, από το Ίδρυμα Αναλύτ, το οποίο είναι υπέρ του πολιτιστικού κοινωνικού διαλόγου. Έχουμε την κυρία Ζαμπίνα Σαούτη, η κυρία Μαρία Φατίνα από την Πορτογαλία. Σωστά το όνομά ε, Ο κύριος Αμπτελουάτ Μαχάπς από το Μαρόκο και η κυρία Καταρίνα Φερασνιέβετς από την Πορτογαλία. Κύριος ε, Σάμια από την Γαλλία. Ε, έχετε συνολικά 15 λεπτά χρόνο να παρουσιάσετε το πρόγραμμα και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου που θα θέλουν να λάβουν πληροφορίες για το πρόγραμμα και να κάνουν ένα διάλογο μαζί σας. Ξεκινάω ε, από σας, ε, κυρία Σαουντή, έχετε το λόγο. Γεια σας. Είμαι η Σαμπρίνα Σαουντή, είμαι manager στο Ίδρυμα Αναλίντ. Έχουμε 42 χώρες. Το Ίδρυμά μας είναι το μεγαλύτερο και το πιο ποικιλόμορφο δίκτυο οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών θέλουμε να προωθήσουμε το διαπολιτισμικό διάλογο στην περιοχή της, ε, την Ευρωμεσογειακή, το Ίδρυμα έχει, παίζει στρατηγικό ρόλο στο διάλογο των νέων σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως με το ρόλο που παίζει ως συντονιστής των, ε, το προγράμματος για τη φωνή των νέων και είναι μέλος για, στο Erasmus Plus και για την εικονική ανταλλαγή. Το πρόγραμμα για τις νέες ευρωπαϊκές φωνές θέλει να αναπτύξει δεξιότητες και δυνατότητες για συζήτηση των νέων στην ευρωμεσογειακή περιοχή και θέλει να υποστηρίξουμε τους νέους να μπορέσουν να μιλήσουν και να εισακουστούν. Η Καταρίνα Ενσαμίρ εδώ θα αναπτύξει την εμπειρία που έχει αποκομίσει ως εκπρόσωπος του Young NetMed Delegate. Το Ίδρυμα Αναλίν ε, προσπαθεί να προωθήσει την κινητικότητα της κοινωνίας των πολιτών και των φοιτητών μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Ε, κάνουμε διαγωνισμούς για κινητικότητα των νέων και με εικονική ανταλλαγή και συζητήσεις. Γι' αυτό το Ίδρυμα ε, η Πορτογαλική Αντιπροσωπεία υποστηρίζει το έρασμος των διαφόρων ενώσεως για να έχουμε ανταλλαγή πολιτισμικών εκδηλώσεων. Και οι συνάδελφοι από την Πορτογαλία και το Μαρόκο θα αναπτύξουν περαιτέρω τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Να τονίσω ότι ετοιμάζουμε εκδηλώσεις. Τέταρτο φόρουμ το Μεσογειακό που διοργανώνεται στα πλαίσια της κρατικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει χώρα στο Σίμπενιτς από 2 μέχρι 5 Απριλίου του 2020. Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 42 κράτη-μέλη της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ένωσης νέων, περιφερειακά ιδρύματα, φορείς ΜΜΕ και διάφορα άλλα ιδρύματα δωρητών και θα εντοπίσουμε προτεραιότητες για την προώθηση διαπολιτισμικού διαλόγου στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά θα έχουμε εκδήλωση υψηλού επίπεδου των νέων ε, της Μεσογείου ε, τον Ιούνιο του 2020. Διάφορες εκδηλώσεις θα διοργανώσουμε. Η συνάδελφος θα αναφερθεί στο, στα διάφορα προγράμματα. Ο κύριος Μαρμπρούρ, ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να παρουσιάσω από πλευρά της ομάδας μου αυτό το όλο πρόγραμμα με τον τίτλο έρασμος των ενώσεων για την πολιτισμικότητα. ΕΡ είναι το ακρονίμιο. Θέλουμε να συμβολήσουμε τη φιλία, την ανοιχτή προσέγγιση προς τον άλλον. Ένα πρόγραμμα είναι αυτό, με στόχο γενικό να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων κινητικότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων και των δύο ακτών του Βορρά και του Νότου, επιτρέπει και κινητικότητα κάθετη μεταξύ Βορρά και Νότου και Νότου και Βορρά, επιτρέπει και μια κινητικότητα μεταξύ των χωρών του Νότου. Και είναι το ισχυρό σημείο ε, του όλου αυτού προγράμματος. Θα δώσω το λόγο την καθηγήτρια Φατίμα να μιλήσει για τι ιδιαιτερότητε και μετά θα μιλήσω εγώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλες και όλους. Εκπροσωπώ την κοινωνία των πολιτών της Πορτογαλίας. Μαζί με το Ίδρυμα Αναλίντ κάνουμε αυτή την προσπάθεια για την κινητικότητα μεταξύ του Βορρά και του Νότου, Βορείου Ευρώπης και του Νότου. Η πρωτοτυπία είναι ότι καλύπτουμε και τις δύο ακτές του Βορρά και του Νότου της Μεσογείου και έχει διτή διάσταση. Πανεπιστήμιο, περιβάλλον και έχουμε και μια άλλη διάσταση κοινωνικο-οικονομική. Η πανεπιστημιακή διάσταση είναι διαπολιτισμική διάσταση, εκολαπτήρια επιχειρήσεων, βιώσιμη ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, απασχολησιμότητα και το Fab Έχουμε σε κοινωνικό επίπεδο προσέγγιση, σημαντικότατη για μας, σημαντικότερη ίσως από το πανεπιστημιακό επίπεδο. Θέλουμε να ανοιχτούμε προς την, στους συλλογικούς φορείς, τις διάφορες ενώσεις σε τοπικό επίπεδο, την κοινωνία των πολιτών, τα τοπικά συμβούλια, επαρχιακά, περιφερειακά, τις ε, διαφόρες ενώσεις των συνεταιρισμών, αθλητικούς συνδέσμους. Έχουμε σαν εταίρους ήδη πολιτισμικές ενώσεις, πολιτιστικές ενώσεις, αθλητικές ενώσεις, πολύ σημαντικό αυτό, και συμμετοχική, συμπεριληπτική είναι η προσέγγιση και στους πτυχιούχους, τους νέους είμαστε ανοιχτοί, αλλά κυρίως στους μη πτυχιούχους. Και αυτό είναι σημαντικό. Μιλάμε η κινητικότητα βορρά-νότου, νότου-βορρά και νότου-νότου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνω με την ανεπίσημη εκπαίδευση, βιοτεχνία, αθλητισμός, νέα επαγγέλματα, λέξεις κλειδιά του προγράμματος. Και ο συνάδελφος το Μαρόκο θα συνεχίσει να περιοριστώ εγώ σε τρεις άξονες. Θα περιοριστώ στον άξονα της, ε, το βιοτεχνικό και εντάσσομαι σε εθνικό πρόγραμμα ένα εργοτάξιο του Μαρόκου με στόχο την τόνωση του τομέα σαν κοινωνικό και οικονομικό φορέα, να έχουμε μια δίκηση με στατηγικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη, να εξασφαλίζουμε επίσης την υποπτία και την πλαισίωση, να ενθαρρύνουμε την ισότητα μεταξύ των φύλων, η ισονομία και αυτονόμηση των γυναικών. Πολλές πτυχές έχουν συμπεριληφθεί. Έχουμε την πτυχή την παραγωγική, η βελτίωση της τεχνικής παραγωγής, εμπορευματοποίηση, να εντάξουμε τους χώρους εμπορευματοποίησης εντός των νέων χώρων για τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη, προώθηση, διαφήμιση, ε, υποστήριξη σε διάφορες εκθέσεις, κατάρτιση, να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα της κατάρτισης με τη βοήθεια εταίρων, Βελτίωση επίσης αυτήν την άλλη πτυχή των συνθηκών διαβίωσης ε, των βιοτεχνών, ανδρών και γυναικών, υγιεινή, ασφάλεια, κάλυψη οικονομική, ποιότητα και τυποποίηση, πιστοποίηση, παραδείγματο χάρη, όσον αφορά την κετοθεσία, καινοτομία και έρευνα σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια πιο συγκεκριμένα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο το σπίτι ε, του βιοτέχνη είναι ένας χώρος ε, για ένα μόνο επάγγελμα, μόνο εργασία, να πλησιάσουμε κυρίως τις γυναίκες. Ε, η ύφανση ε, χαλιών, εκθέσεις, εμπορευματοποίηση των βιοτεχνικών προϊόντων. Θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας, κυρίως για την προστασία των γυναικών και θέλουμε να βοηθήσουμε με εργαλεία παραγωγής. Όλος μηχανισμός φαίνεται εδώ, στο διάγραμμα, δίκτυο σε εθνικό επίπεδο, κάλυψη παρέχεται, όλης της επικράτειας των περιοχών του Μαρόκου, μπορούμε να υποδεχτούμε σχεδόν 14.000 άτομα, πρακτική κατάρτιση και θεωρητική λαμβάνει η χώρα, Βλέπετε εδώ οικονομική προσέγγιση που καλύπτει και την ε, κινητικότητα βορρά-νότου-νότου-βορρά και νότου-νότου. Μετά βασιζόμαστε σε συμπράξεις και συνεργασίες ευρείες πανεπιστημιακό επίπεδο με από πανεπιστήμια του Μαγκρέμπ αλλά στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Πορτογαλία κλπ και διάφορες ενώσεις και συνδέσμους και θεσμούς που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα που προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη και έχουμε κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους εδώ διάφορους φορείς εθνικούς και στην Αλγερία και στην Τινησία και στην Πορτογαλία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, με λένε Κατερίνα Νέβες και είμαι 24 ετών, είμαι από την Πορτογαλία και ανέκαθεν θεωρούσα τον εαυτό μου ως Ευρωπαίο πολίτη. Είμαι Ευρωπαία και μετά από τις εμπειρίες που πραγματικά ε, προσδιορίσαν την ταυτότητά μου, μπορώ να πω ότι νιώθω και μεσόγεια, μεσογειακή. Έχω συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο για την ηγεσία τον Ιανουάριο πέρσι ε, στη Μάλτα. Εκεί συναντήθηκα με τον καλό μου φίλο τον Σαμίρ και τα υπόλοιπα μέλη της μεσογειακής οικογένειας. Το πρόγραμμα YMV δίνει σε νέους και από τις δύο όχθες της Μεσογείου διάφορες δεξιότητες για την ηγησία, για την ερητορία, για, την, ε, για το δημόσιο διάλογο, δεξιότητες που τους χρειάζονται στις συναλλαγές τους και στη συνύπαρξη και την επικοινωνία με τους ηθήνοντες για τη χάραξη της πολιτικής, με τους δημοσιογράφους, με εκπροσώπους των ΜΜΕ, δεξιότητες πολύ σημαντικές. Έχουμε 5 συν 5 Υπουργική διάσκεψη 5 συν 5 ε, στο πλαίσιο του YMVI και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με αυτούς τους επικεφαλείς, ε, τους πολιτικούς, για την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι νέοι στη διαδικασία λήψης απόφασης και για στη διαδικασία για τη σφαιριλάτηση της μεσογειακής ταυτότητας. Ο Υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, ο Κουστίν Σίλβα, με ε, προσκάλεσε να συμμετάσχω σε μια αντιπροσωπεία η οποία θα συμμετείχε σε διάφορα φόρουμ σχετικά με το θέμα αυτό. Κατά, καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία, αυτό το οποίο με εντυπωσίασε είναι το εξή. Όσο και αν γίνεται λόγο για το μέλλον και για του νέου. τελικά η φωνή των νέων δεν ακούστηκε ιδιαίτερα. Δεν ήταν πολλοί οι νέοι που μπόρεσαν να κάνουν τη φωνή του να ακουστεί καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία. Έτσι και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την κινητικότητα των νέων και τη συμμετοχή των νέων. Τώρα, να σα πω κάτι πιο προσωπικό. Η κινητικότητα είναι αυτή που διαμόρφωσε και την προσωπικότητά μου. Ε, αυτή που με έκανε Ευρωπαία πολίτη και ε, νιώθοντας επίσης και μεσογειακή. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα κινητικότητας, ανταλλαγές σπουδαστικές, ε, προγράμματα εκπαίδευση. Με το πρόγραμμα Εράσμου αναπτύχθηκα προσωπικά και κοινωνικά και θέλω και άλλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως αυτές που είχα εγώ. Και γι' αυτό αυτό το project, το Εράσμου των Συλλόγων και των Ενώσεων, είναι πολύ σημαντικό γιατί λειτουργεί συμπεριληπτικά. Νέοι από ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε, από την Ήπεθρο επίση, από απομακρυσμένε γεωγραφικέ περιοχέ, μπορούν να αξιοποιήσουν, να δρέψουν τα ωφέλη τη κοινωτικότητα των νέων. Για να δώσουμε τη δυνατότητα στου νέου να αποκτήσουν τι ικανότητε, να χαράξουν πολιτική αύριο, πρέπει να του δείξουμε, αλλά και κυρίω πώ γίνεται, αλλά και να του επιτρέψουμε να αναλάβουν αυτό το ρόλο τη χάραξη πολιτική αύριο. Βοηθήστε λοιπόν να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σα. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ τι εμπειρίε μου ε, για την κοινοτικότητα. Με λένε Σαμίρα Κασά, είμαι 32. Όταν ήμουν μικρό, έφυγα από την Αλγερία το 1995 με την οικογένειά μου για να ξεφύγω από την τρομοκρατία. Έχασα την αγάπη τη ζωή μου. Φαντάζεστε πόσο φοβερό ήταν αυτό για ένα 7χρονο παιδί. Ε, πιο μετά μπορεί και να ξαναβρεθήκαμε στο facebook, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλη ιστορία. Στη Γαλλία εντάχθηκα γρήγορα, καταβρόχθησα τα βιβλία, προσπαθούσα να μάθω όσο γρήγορα γίνεται. Ε, ε, η διηγητική μου γειτονιά δεν, ήταν, δεν είχε καθόλου ποικιλομορφία. Ε, ήμασταν όλοι περισσότεροι μαύροι Άραβες. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχα π.χ. γνωρίσει κανένα Εβραίο και δεν είχα Εβραίο φίλο. Στο Πανεπιστήμιο σπούδασα πολλά και διαφορετικά πράγματα για τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνο άλλαζα βασικό πτυχίο και τελικά τα παράτησα. Οι γονεί μου θυσίασαν τα πάντα αλτροιστικά για να έχουμε εμεί ένα καλύτερο μέλλον και πίστευαν ότι το πανεπιστήμιο είναι ο μόνο τρόπο να πάμε μπροστά. Ε, τα παράτησα από το πανεπιστήμιο και για έξι μήνε έπαιζα ένα βιντεοπαιχνίδι, το Second Life. Έτσι έμαθα καλά αγγλικά και τελικά έβαλα στο Google τι να κάνω με τη ζωή μου. Και ε, ανακάλυψα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού. Συμμετείχα. Μου άρεσε πάρα πολύ να παίρνω φωτογραφίες και βίντεο, ενώ δεν έχω ιδιαίτερα προσόντα. Το γραφείο λοιπόν αυτό μου έδωσε μια φωτογραφική μηχανή και μου έδωσε την ευκαιρία να βιώσω ε, την εμπειρία που θα ήθελα. Οργανώσαμε ένα debate, μια συζήτηση για την άκτα και καλέσαμε τρία πολιτικά ε, κόμματα, τρεις πολιτικές ομάδες από το κίνημα Occupy. Και τελικά ε, είχαμε και συνάντηση στα Σουηδικά χωρίς να καταλαβαίνω λέξη. Επέστρεψα στην ε, Γαλλία και ένιωσα ότι έχω πολύ μεγάλη ικανότητα. Ένιωσα ότι ε, είχα δυνατότητα, μπορούσα να κάνω. Με το Erasmus Plus ταξίδεψα και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ταξίδεψα και στην Ιερουσαλήμ στη συνέχεια και πήρα μέρος στο διαθρησκιακό διάλογο. Σας είπα νωρίτερα ότι δεν είχα ποτέ Εβραίο φίλο. Με προσκάλεσαν στη συναγωγή. Ε, και όταν έφυγα από το σπίτι μου, λέω, ε, είπα στον εαυτό μου πώς θα πάω στη συναγωγή. Έχω ξεχάσει το κυπά, το ε, καπελάκι των Εβραίων. Στη συνέχεια όμως τους ε, ε, τους ε, ε, φιλοξένησα και εγώ και τους κάλεσα στο ΑΕΤ στη δική μας θρησκευτική ζωή και γιορτή και είχαμε την ευκαιρία να φάμε κουσκούς στα παραδοσιακά μας φαγητά. 30 μήνες ταξίδευσα σε όλο τον κόσμο και καταγράφω σε ηχητικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό το διαθρησκιακό διάλογο με, την, ε, με το Ίδρυμα Αναλίντε έχω έρθει πάλι σε σύνδεση με τις αραβικές μου ρίζες και θέλω να δουλέψω για το, το, το στόχο, ε, τους στόχους ε, της αηφόρου ανάπτυξης. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για όλη αυτή τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σφυριλάτηση της δικής μου ταυτότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις σας που μας εισάγουν στο έργο σας ήταν και μαρτυρίες ταυτόχρονα. Είναι πολύ σημαντικό ε, κανείς ε, να μπορεί να βλέπει έτσι πιο βαθιά πώς ε, βιώνουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα. Ανοίγω λοιπόν τη συζήτηση και οι βουλευτές μας έχουν τον λόγο. Η κυρία Στράτοβα έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που θέλουμε να υποστηρίξουμε το Εράσμους ως πρόγραμμα να διευρύνουμε τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουμε να γίνει πιο μαζικό το πρόγραμμα και να μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αυτό. Έχω μια ερώτηση για σας, γιατί μάλλον δεν το σημείωσα, δεν το κατάλαβα. Από την παρουσίασή σας βλέπω ότι το project είναι αρκετά μεγάλο. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός, για πόσα χρόνια, ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και πόσοι. Θα ήθελα να ξέρω γιατί βλέπω ότι είναι ένα έτσι πολύπλευρο και μεγάλο σχέδιο. Θα ήθελα μια εικόνα σχετικά με τον προϋπολογισμό και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να μαζέψουμε τις ερωτήσεις και μετά να έχουμε μια συνολική απάντηση. κυρία Πέτρα Καμαέβερτ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή του σχεδίου, αυτού του έργου που είναι πραγματικά συναρπαστικό. Βλέπω ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου μπόρεσαν να έχουν μια καλή σύνδεση μεταξύ τους και πραγματικά μου αρέσει το γεγονός ότι επικεντρωθήκατε όχι μόνο στον ακαδημαϊκό κλάδο, αλλά και στο μη ακαδημαϊκό. Μιλάμε για συγκεκριμένες σχέσεις, ε, για την βιοτεχνία, ε, για νέες μορφές ε, βιοτεχνικής εργασίας. Επίσης για το όνομα, να είμαι λίγο ειλικρινής, δεν μου αρέσει καθόλου να χρησιμοποιείται έτσι πλεονασματικά ο όρος Εράσμους, γιατί κανείς τελικά δεν γνωρίζει για τι μιλάμε. Εράσμους είναι το μεγάλο πρόγραμμα κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς μεταξύ μας έχουμε συχνά την τάση και από την πλευρά της Κομισιόν να λέμε ένα «εράσμος» για το τάδε ή το δίνα ε, για τους ε, καλλιτέχνες π.χ. Στο τέλος, κανείς δεν ξέρει γιατί μιλάμε. Είναι το Εράσμος ή κάτι καινούριο. Γι' αυτό λίγο με πειράζει αυτή η πλεονασματική χρήση της ε, έκφρασης αυτής. Καλό είναι να έχουμε μια καθαρότητα στα ονόματα και να μην ε, ε, ε, έχουμε έτσι μια συγκεχημένη άποψη ε, για το τι μιλάμε, γιατί έτσι χάνει και την αξία του λίγο. Έτσι, δι, λίγο το θέμα και δεν ε, έχει την ίδια αξία. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Oh, Ευχαριστώ. Εγώ Χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που σας ε, υποθέχομαι για πολλούς λόγους σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού εντός της αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ενώσεως για τη Μεσόγειο είχα ζητήσει, είχα εκφράσει την ευχή να οικοδομήσουμε ένα έρασμο σε όλες τις ε, χώρες ε, της Νοτιού Μεσογείου, ένα ισχυρό έρασμος, όπως αυτό που γίνεται στην, στο Μαρόκο, να έχουμε συμπεριληπτικό πλαίσιο, να προχωρήσουμε πιο πέρα τα πανεπιστήμια με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα για να απαντήσω στον κύριο Λυσμόνης το όνομά σας. Με συγχωρείτε και δεν βλέπω. Μετά τα 40 δύσκολο να βλέπει κανείς τόσο μακριά βλέπετε. Α, ευχαριστώ. Τι πλούτο μπορεί να δώσει η διαπολιτισμικότητα και εγώ με ένα τέτοιο προϊόν διότι είχα γαλλική παιδεία, γεννήθηκα στη Γαλλία και αλγερινή εκπαίδευση διότι είναι αλγερινή γονείς μου με έχουν εμπλουτίσει οι δύο αυτοί πολιτισμοί και το διατυμπανίζω θα πρέπει να εκμετατευτούμε τον πολιτικό, πολιτισμικό πλούτο των χωρών της Μεσογείου σε κάθε ευκαιρία εγώ θέλω πράγματι να συνεργαστούμε στα πλαίσια του έρασμος, διότι είμαι και σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας μου και σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κουλτ της Euromed το θέλω αυτό. Σας περιμένω, θα συνεργαστούμε και σας ευχαριστώ για αυτά τα όμορφα προγράμματα που εφαρμόστε. Η κυρία Λίγο να έχουμε πρώτα μια απάντηση, αν είναι εύκολο. Σα ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε αυτά τα όμορφα προγράμματα. Είχα μια ερώτηση που αφορούσε και την προηγούμενη. Το επίπεδο τη κινητικότητας, διότι ο Erasmus ΣΥΝ είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας. Έχετε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα πολύ για τη βιοτεχνία. Το σε αυτό. αλλά πού εντασσόταν η διάσταση της κινητικότητας. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις παρακαλώ. Άλλη ερώτηση. Μίλησατε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εκπαίδευση τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των προγραμμάτων. Συζητάμε το θέμα της παιδείας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Γι' αυτό θα με ενδιαφέρει να μου πείτε ποια είναι η εμπειρία σας. Πώς εφαρμόζετε, υλοποιείτε αυτού του είδους τα προγράμματα. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε με την απάντηση. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας σας πρώτα απ' όλα για τις ερωτήσεις που είχα την καλοσύνη να μου θέσατε για τον προπολογισμό. Περίπου καμία εκατοστή κινητικότητα στο χρόνο από βορρά προς νότο, νότο βορρά και σε οριζόντιο επίπεδο κινητικότητα. Ενδεικτικά είναι τα νούμερα που αναφέρουμε θα πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειες κινητικότητας κατά 100 το χρόνο. Μπορούμε να καλύψουμε έτσι την κινητικότητα και να διαχειριστούμε την κινητικότητα. Με τη βοήθεια των εταίρων και του Βορρά και του Νότου και τη βοήθεια των κοινωνικο-οικονομικών εταίρων των διαφόρων συνδέσμων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και των ενώσεων. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, η κινητικότητα αφορά τους πτυχιούχους και τους μη πτυχιούχους. Ο όρος έρασμος είναι ε, ιερός όρος. Ο καθένας καταλαβαίνει, ένα συγκεκριμένος όρος. Ο, κα, καθένας καταλαβαίνει περί πρόκειται. Έχουμε το έρασμος, το έρασμο συν, Όλος ο κόσμος γνωρίζει το Εράσμος είναι ένας παράγων ένωσης των νέων της Ευρώπης, των νέων φοιτητών στα πανεπιστήμια. Είναι ένα πρόγραμμα κινητικότητας ευρύτερο, μεγαλύτερο από την κινητικότητα Εράσμος, αυτό που συζητάμε, διότι αφορά και άλλα μέλη του κοινού, το διαφορετικό κοινό, από, κοινωνικ... από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όχι μόνο τους φοιτητές των πανεπιστημίων, κυρίως τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή παιδεία και την ανώτατη παιδεία. Να πάμε λίγο σύντομα. Καταρχάς να πω ότι το Erasmus Plus δεν είναι Erasmus. Το Erasmus ήταν καθαρά για τους ε, φοιτητέ. Το Erasmus Plus είναι για την επαγγελματική εκπαίδευση, για την ανταλλαγή δασκάλων, ε, μαθητών. Δεν είναι μόνο ακαδημαϊκή. Το Erasmus ε, Plus έχει να κάνει με τις επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα και δεν είναι μόνο για τους φοιτητές. Αυτό ήθελα να το διευκρινίσω και εγώ να επανέλθω σε κάτι που θίξατε. Προφανώς θα επιμείνουμε επί της κινητικότητας, της διαπολιτισμικότητας. Η πρωτοτυπία του προγράμματος είναι ότι θα επιμείνουμε κατά πολύ στον πολιτισμικό τομέα, τη βιοτεχνία, τον αθλητισμό. Είναι κάτι καινοτόμο, κάτι που ξεπερνά το Erasmus Αυτό το παρόν ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα χαρώ να έρθω σε επαφή μαζί σας, να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το όλο πρόγραμμα. Όσον αφορά τα οικονομικά, γεννήθηκε με τη Σύνοδο Κορυφής των δύο ακτών της Μεσογείου. Έχουμε σε επαφή με τα κάτι μέρη που μας υποστηρίζουν και έχουμε ιδιωτικού πόρους, ειδικού πόρους για την κινητικότητα που μας στηρίζουν οικονομικά Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα με ένα χρονοδιάγραμμα για να εντοπίσουμε τους δικαιούχους νέους μέχρι το τέλος του έτους. Το Ίδρυμα Άννα με 42 χώρες που συμμετέχουν. Μεταξύ ε, ε αυτών έχουμε 4.600 με 5.000 ενώσεις. Έχουμε μία βάση συνδέσμων και ενώσεων για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και τα διάφορα στοιχεία και να αναπτύξουμε συνεργασία με αυτές τις ενός και τους συνδέσμους. Να επανέλθω στη σχέση μεταξύ παιδείας και βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ίδρυμα Αναλίντ. όλο και περισσότερο κινείται μέσω των Intercultural Trend Reports, των εκθέσεων αυτών και βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις στην παιδεία και συσχετισμός παιδείας και βιώσιμης ανάπτυξης. Όλο και περισσότερο συνεργαζόμαστε με τους νέους, με τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης και κάνουμε πάρα πολλή δουλειά με αυτούς τους νέους προσπαθώντας να συνδέσουμε τα διάφορα σημεία, τα διάφορα στοιχεία με τα χαράς να τα συζητήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω μαζί αυτά τα στοιχεία. Όσον αφορά το, τη βιοτεχνία, πριν από αυτό. Το ερώτημα της κυρίας Αντιπροέδρου. Α, έφυγε. Την κινητικότητα το άνοιγμα που δεν αφορά μόνο τον πανεπιστημιακό κόσμο. Το είπαμε και στην παρουσίαση. Έχουμε ανοιχθεί λοιπόν προς τις, ε, στους διάφορους συνδέσμους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς και στην τοπική οργάνωση και αυτοδίκηση. ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι όλοι αυτοί οι φορείς να συμμετέχουν στις δράσεις μας. Η κινητικότητα και ο τεχνικός κλάδος Πώς εξηγούμε την κινητικότητα βορρά-νότου κυρίως. Αν μιλήσω για το Μαρόκο, είναι γνωστή βιοτεχνία του Μαρόκου και υπάρχουν πολλοί μαθητευόμενοι στην Ευρώπη που θα ήθελα μια τέτοια εκπαίδευση σε αυτό το πλαίσιο. Εντός των διαφόρων φορέων που βρίσκονται στο Μαρόκο και αυτό θα είναι υπεραξία όσον αφορά τη χρησιμότητα, αλλά και για να γνωρίζουν οι μεν τους δε, ο ένας τον άλλον. Το να δέχεται ο ένας τον άλλον, κάτι που επιδιώκουμε σαν στόχο. Συμπροματικές πληροφορίες για την κινητικότητα νότου-νότου. Δύο παραδείγματα έχω. Τι ζήσαμε στα πλαίσια της έρευνας. Το PHC, έχουμε ε, ε, συνεργασία Αλγερίας, Τινησίας, Μαρόκου με γαλλικά εργαστήρια. Λειτουργήσε πολύ καλά το πρόγραμμα. Πέρα από την κινητικότητα βορρά-νότου-νότου-βορρά, επέτρεψε κινητικότητα και συνεργασία νότου-νότου και εκεί έχουμε δίκτυο νέων ερευνητών. οι οποίοι στις έρευνές του συνεργάζονται, ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα και έχουμε και ένα κολέγιο για διδακτορικά στο Μαγκρέμπ, 27 μεταπτυχιακούς φοιτητέ. έχουμε εκεί από Μαρόκο, Αλγερία, την Ισία, Βέλγη, συμμετοχή Βέλγων και Γάλλων. Παρακολουθήθηκαν επί τριετία, δημιούργησαν ένα δίκτυο ερευνητών. Δίκτυο που θα μπορούσε να λειτουργήσει, να είναι επιχειρησιακό, λειτουργικό τα επόμενα χρόνια. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πέτρα Κάμα Έβερτ. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω ότι είναι εξαιρετικό αυτό το πρόγραμμα. Μόνο το όνομα λίγο με ενόχλησε γιατί φοβήθηκα ότι χρησιμοποιείται το όνομα Εράσμους έτσι πλεονασματικά όπως είπα και στο τέλος χάνει το βάρος του. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το έργο είναι καλό. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είναι όμως τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε στην Ευρώπη. Έχω και μία ερώτηση. Περιμένετε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να το κάνετε πιλωτικό πρόγραμμα. Ή λέτε εμείς τα καταφέρνουμε με τους εταίρους μας, ε, αυτούς που έχουμε δηλαδή στο Ίδρυμα και τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Και εγώ έχω μια επερώτηση. Το δικό μας ε, πρόγραμμα είναι ε, περιορισμένο σε συγκεκριμένες χώρες, εκτός από το Erasmus Mundus φυσικά. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε ε, επικεντρωθεί και στην εταιρική σχέση βορρά-νότου. Ε, θα ήταν, αν το κάναμε αυτό, θα ήταν μια επέκταση του ευρωπαϊκού προγράμματος. Αυτό που ρώτησε ήδη και η Πέτρα είναι σημαντικό Πώς είναι η χρηματοδότηση του Ιδρύματος, τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς χρηματοδοτείτε το Ίδρυμα, έχετε τα δικά σας μέσα ως Ίδρυμα, αλλά ε, πώς χρηματοδοτήσατε ε, τα προγράμματά σας και τις ιδέες σας ως τώρα. Περιμένουμε από σας μια απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι. Ελπίζουμε και μπορεί Ελπίζουμε να δούμε πώς θα τα αναπτύξουμε όλα αυτά με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής ε- Ένωσης. Ίσως το δούμε αυτό αργότερα με την Αντιπρόεδρό σας, με ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Για τα σχέδια, τα έργα και τις δραστηριότητές μας σε γενικές γραμμές έχουμε οικονομική στήριξη ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους περίπου 70% ε, αλλά και στήριξη από τα κράτη-μέλη. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όντως, Έχουμε προς το παρόν στήριξη από τον ιδιωτικό τομέα, ο Απτελουαχέτε μας το υπενθύμησε, και προς το παρόν πορευόμαστε έτσι, με τη στήριξη ιδιωτών. Ελπίζουμε να έχουμε πολιτική στήριξη από το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το ξεκινήσουμε ως πιλωτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Από την πλευρά σας υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ, κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτού του προγράμματος. Ε, να πω, ομολογώ ότι δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η στόχοθεσία, η κατεύθυνση του προγραμματός σας. Ε, έχω κάποιες ε, πληροφορίες, αλλά δεν με διαφωτίζουν ιδιαίτερα. Έχω ένα ερώτημα. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή την Επιτροπή ε, έχει συμμετοχή 70%. 70% από ποιο ποσό. Πόσα έχετε στη διάθεσή σας. Και είπατε ότι το Μαρόκο δίνει, ε, ε, θα έχει ένα ίδρυμα, όμως για την εκπαίδευση συγκεκριμένα. Όμως μετά από αυτή την εκπαίδευση ποιες ε, θα είναι οι προοπτικές εργασίας. Συγκεκριμένα στην αγορά εργασίας ε, ποια είναι τα δεδομένα ε, και αν αξίζει τον κόπο αυτή η προσπάθεια. κυρία Σαουντή, όταν μίλησα για το 70% εννοούσα για τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Αναλίντ κατά 70%, αλλά ίσως έχετε εσείς περισσότερα στοιχεία για το άλλο ερώτημα να απαντήσετε. Ο κύριος Μαρμπρούρ. Ε, σας ευχαριστώ, κυρία Βουλευτή. Το παράδειγμα αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων. Το σπίτι του οικοτέχνη ή βιοτέχνη είναι ε, σπίτια, είναι οίκοι, είναι ιδρύματα που μπορούν να υποδεχθούν νέους από τον Νότο ή από το Βορρά για να τους προσφέρουν κατάρτιση ή συμπληρωματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Προς το παρόν είναι ιδρύματα αυτά που αφορούν μόνο τους νέους Μαροκινούς που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές ή σε κάπως πιο δύσκολες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για εκπαιδευτικά ιδρύματα, για κέντρα κατάρτισης που μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες τους σε ασκούμενους, σε νέους από την Ευρώπη, από την Τινησία, από το Μαρόκο, για να συμπληρώσουν την ε, κατάρτισή τους για τη χύψη ε, δεξιότητα. Τώρα, ως προς το δεύτερο ερώτημα... Α, συγγνώμη. Αυτό λοιπόν έλεγα είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν τρει άξονε. Πρώτον, η οικοτεχνία, βιοτεχνία. Δεύτερον, το πολιτιστικό σκέλο. Και τρίτον, τα αθλήματα. Θα δουλέψουμε πάνω στου τρει πυλώνε. Ε, αυτό για την οικοτεχνία και τη βιοτεχνία είναι ένα παράδειγμα. Έχουμε αντίστοιχα ε, ίδια παραδείγματα, πολιτιστικά ιδρύματα, καλλιτεχνικά ιδρύματα, αλλά και αθλητικά κέντρα και μπορούν να υποδεχθούν νέου και από το βορρά και από τον νότο. Είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων. Δεν ξέρω σας απάντησα, ελπίζω ναι. Ναι, να κάνω και μια ερώτηση στην Κομισιόν. Τα χρήματα που δίνονται στο Ίδρυμα αναλύνται από πού προέρχονται, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, είναι από την ανάπτυξη, από ποιον κορβανά βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Μπορεί η Κομισιόν να μας πει κάτι σχετικά με αυτό. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να πω ότι δεν το ξέρω. Δεν είναι από τη Γενική Διεύθυνση έργα. Είναι από τα εξωτερικά κονδυλία. Θα το ψάξω και θα το μάθω. Εκτός και αν ξέρει ο εκπρόσωπος από το Ίδρυμα Αναλίν και μπορεί να απαντήσει ήδη αυτό το ερώτημα. Ή εκπρόσωπος. Ναι, η κυρία Σάουντι. Ναι, θα θέλουμε τη στήριξή σας. Θέλουμε τη στήριξή σας. Είναι πολύ χρήσιμη. Wie gesagt, Development ε, αν είναι από την ανάπτυξη ή από την ε, υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης, θα έχει να κάνει με τη συνεργασία με μη ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα είναι πρόγραμμα Εράσμους. Εμείς εδώ ως Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε θέσει μεγάλη έμφαση ακριβώς στο πώς η εξωτερική μας πολιτική μπορεί να βοηθηθεί αν δώσουμε αξία στην εκπαίδευση, και ε, την ε, κατάρτιση, να έχουμε καλύτερες προοπτικές δηλαδή για τους νέους. Αυτό είναι ένας από τους στόχους ε, της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ανάπτυξης. Το Ίδρυμα Αναλίντ στην ουσία λίγο πολύ απευθύνεται στις χώρες της Βορείου Αφρικής, τις ενεργοποιεί και συνεργάζεται μαζί τους ε, για να υπάρχει μια ανταλλαγή, ένας διαπολιτισμικός διάλογος. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ καλό ε, να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και αν γίνεται κάτι χωρίς δικά μας χρηματοδοτικά μέσα, αλλά από την εξωτερική υπηρεσία δράσης, ε, εξωτερικής δράσης, ε, τότε ακόμα καλύτερα. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Αναλίντ για την παρουσία τους εδώ σήμερα είναι εξαιρετικά τα προγράμματά σας, ε, μας πάνε ένα βήμα παραπέρα και πραγματικά μακάρι και με άλλους τρόπους να μπορούσαμε να βοηθούμε τους ανθρώπους στην καθημερινή του ζωή, στην εκπαίδευσή τους. Ε, καλό είναι να μπορούμε να έχουμε τέτοιες παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, έχουμε σήμερα ένα έτσι ε, πυκνό πρόγραμμα σχετικά με τις ακροάσεις, ε, παρουσιάσεις. Τώρα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Το Φόρουμ Νεολαίας λοιπόν είναι ο φιλοξενούμενός μας σήμερα. Ε, πέρυσι το Νοέμβρη ξεκινήσαμε μια προσπάθεια την οποία συνεχίζουμε συγκεκριμένα για την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα νεολαία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φρανσουά Μπαλάτ που είναι Διευθυντής ε, Πολιτικής και Advocacy. Policy Officer επίσης έχουμε την κυρία Τσασίκα που είναι επίσης στο ίδιο θέμα υπεύθυνη και θα έχουμε μία παρουσίαση για το θέμα της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Η κυρία Καμέβερτ και οι, συντονισμοί, και οι συντονιστές ε, είπανε, όρισαν την ε, πρωτεύουσα την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας ε, για το 2020 και Θέλουν να οριστεί η εντολή της ε, πρωτεύουσα αυτής, ε, θέλουμε να υπάρξει μία συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώς ακριβώς θα υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά και μετά θα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση με τους βουλευτές. Ε, ποιος ξεκινάει? Ο κύριος Μπαλάντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή που μας δέχεται εδώ σήμερα. Ε, βλέπω ότι ε, για άλλη μία φορά ξεκινάμε όλοι μαζί να χτίζουμε πράγματα. Θα σας μιλήσω σήμερα για ένα από τα μεγάλα project του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Ε, είχαμε ε, στο παρελθόν μιλήσει για, το ευρωπαϊκό, για την ευρωπαϊκή εκδήλωση της νεολαίας. Ε, θα σας δούμε, ελπίζω, το Μάιο, στις 28-29 Μαΐου φέτος σε αυτήν. Εγώ και οι συνάδελφοι θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Νεολαίας. Είναι μια πρωτοβουλία που εδώ και μια δεκαετία ενισχύει τους νέους ε, και τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας τους σε διάφορες ε, πόλεις της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα των Νεολαίας δεν είναι κάποιος τίτλος, έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με το περιβάλλον, την ψηφιακή οικονομία, με πολλούς τομείς. Όμως, ο νέος αυτός τίτλος ε, στην ουσία μας δείχνει ότι πρόκειται για ε, τους νέους, ε, είναι υπέρ των νέων, για τους νέους, ε, από τους νέους και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, ένα ταξίδι που κάνουν οι νέοι όταν η πόλη τους γίνει Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. 2023 θα γίνει η πόλη μας ε, ε, η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Ε, σας καλώ λοιπόν να παρευρεθείτε κατά τη διαδικασία επιλογής των πόλεων. Εμείς συλλέγουμε τις υποψηφιότητες, φτιάχνουμε την επιτροπή που θα επιλέξει τις πόλεις, κάνουμε την ψηφοφορία, αλλά κυρίως ορίζουμε τους βασικούς Στόχου. Ξέχασα να σας δείξω τις διαφάνειε. Συγγνώμη. Δεν είχα μια οπτικοακουστική υποστήριξη. Ποιοι είναι οι στόχοι της πρωτεύουσα. Η συμμετοχή των νέων να είναι δηλαδή στην καρδιά των αποφάσεων στις πόλεις τους, η δημιουργία ενός ισχυρότερου χώρου για την κοινωνία των πολιτών εντός ε, των πόλεων έχει να κάνει δηλαδή με τα δικαιώματα, το δικαίωμα του συνέρχεσθε, της έκφρασης. Ε, επίσης είναι η δημιουργία δεσμών μεταξύ της ε, Ευρώπης και των τοπικών κοινωνιών δεν έχουμε μόνο τους ε, συνήθεις ύποπτους της ε, πολιτικής νεολαίας. Έχουμε ένα mainstreaming. Όλοι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν για την πόλη τους ε, μπορούν να συμμετάσχουν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενσταλάξουμε την αλλαγή. Πάνω από 130 διαφορετικές χώρες από την Ευρώπη έχουν κάνει αίτηση για τον τίτλο αυτό από την αρχή της πρωτοβουλίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μπορεί να έχουμε ένα μικρό αριθμό πρωτεύουσων τελικά, όμως ε, ε, όλες αυτές οι πόλεις κάτι έχουν πετύχει, έχουν ε, ξεκινήσει την αλλαγή στην πόλη τους μέσα από την, τους οργανισμούς τις οργανώσεις των νέων. Και αυτό είναι ένα εντυπωσιακό επιτεύγμα. Έχετε ήδη λάβει υλικό για τη σημερινή μας συνάντηση και μέσα σε αυτό υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. 8.000 πρωτοβουλίες, πάνω από 8.000 εκδηλώσεις, δραστηριότητες της πόλης. Πραγματικά έχει φέρει αλλαγή αυτή η δράση. Σας φέρνουμε εδώ τις μαρτυρίες νέων εθελοντών από τις πόλεις. Όταν κάνουμε συνεντεύξεις με τους νέους, Πραγματικά βλέπουμε ότι πιστεύουν ότι συνέβη αλλαγή στις χώρες τους, στους δήμους τους, σε όλες τις δομές των πόλεων τους. Ε, θεωρούν ότι έχουν μπει στη θέση του οδηγού. Επίσης έχει δημιουργηθεί ένας χώρος για ενεργό συμμετοχή των νέων. Όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες νεολαίας έχουν ε, διαφορετικά μοντέλα, δεν υπάρχει ένα ενιαίο. Ε, ας πούμε έχουν γίνει εργαστήρια δημιουργικότητας. Πώς να έρθουν οι νέοι στο τραπέζι, πώς να συναποφασίζουν για το μέλλον της πόλης τους. στην Επιτροπή Πολιτισμού φυσικά να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και το θέμα των εθελοντών. Πάνω από 10.000 εθελοντές ε, έχουν εμπλακεί σε αυτά τα project ε, αυτό το διάστημα. Δείχνει ακριβώς πόσο χρόνο, πόση αφοσίωση ε, αφιέρωσαν και επένδυσαν σε αυτά τα προγράμματα. Έχουμε επίσης τη δημιουργία ενός στενού συνδέσμου μεταξύ της τοπικής τους ταυτότητας και της ε, εθνικής και ευρωπαϊκής τους ταυτότητας. Ε, στην ουσία έχουμε ε, μία ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της συμμετοχής όλων των ομάδων. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, είχαμε ένα πολύ καλό μοντέλο προς αυτή την κατεύθυνση. Ανέφερα επίσης και την ενίσχυση των οργανώσεων των νεολαίων. Συνολικά ε, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ επένδυσαν οι πόλεις αυτές ε, μέσα σε αυτό το διάστημα σε τέτοια project. Και τέλος να αναφέρω, μίλαγα πριν για την σχέση μεταξύ της τοπικής και της ευρωπαϊκής διάστασης, ε, να πω ότι έχουμε κάθε χρόνο ένα διεθνές σημείο συνάντησης. Οι εκπρόσωποι από τους οργανισμούς νεολαίας σε όλη την Ευρώπη συνέρχονται, συναντιούνται για να συζητήσουν ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις, τι διακυβεύεται σε επίπεδο ε, νεολαίας. Ε, στην πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 θα μιλήσουμε για τη βιωσιμότητα, ε, τη δημοκρατία, ένα φόρουμ δημοκρατίας στην πραγματικότητα δημιουργούμε. Αυτό το project, όπως βλέπετε, έχει πετύχει πολλά τις τελευταίες, ε, την τελευταία δεκαετία και θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα. Είμαι περήφανος πραγματικά για τους συναδέλφους, τη Ρίτα και τους άλλους που έχουν δημιουργήσει αυτό το εξαιρετικό project Αλλά υπάρχουν βασικές ε, προκλήσεις. Καταρχάς, ε, πώς αυξάνουμε την ε, ορατότητα αυτού του στόχου, πώς συνεργαζόμαστε με τους διάφορους εταίρους, πώς φτάνουμε σε επίπεδο ορατότητας, πώς συνεργαζόμαστε. Και από την άλλη, όπως βλέπετε εδώ και στη διαφάνεια, υπάρχουν πράγματα που μπορούν ακόμα να γίνουν σε επίπεδο οικονομικής υποστήριξης, να υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής που θα υποστηρίξει τις πόλεις που θα πρέπει να εργαστούν για μια σειρά ετών για να προετοιμάσουν αυτή τη διαδικασία και δεν θέλουμε αυτά τα project να είναι μόνο ετή, θέλουμε να αφήσουν μια κληρονομιά, να ενσταλάξουν την αλλαγή όπως είπα στις πόλεις. Σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε αυτό το project σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας προσκαλέσατε. Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Στην Επιτροπή Κούλτ. Και όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Νεολαίας. Θέλουμε να διαρευνήσουμε την εταιρική σχέση μεταξύ μας, πιθανές επισκέψεις. Ξέρω ότι πάτε στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Ε, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να κάνουμε και στη δική μας περίπτωση πώς να συνεργαστούμε, πώς η Επιτροπή Πολιτισμού μπορεί να είναι πιο πολύ παρούσα να υποστηρίξει τις πόλεις ε, να δώσει μία σύνδεση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, να υπάρχει μια στενότερη συνεργασία δηλαδή μεταξύ της Επιτροπής και των πόλεων. Ξέρουμε επίσης ότι η Επιτροπή σας υποστηρίζει εξαιρετικά προγράμματα όπως το Erasmus Plus το Ευρώπη των, για τους πολίτες, ε, το Σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα συνδέσουμε με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Νεολαίας, να δημιουργήσουμε hubs, ε, κάποια κομβικά σημεία, στα οποία οι νέοι κάθε χρόνο μπορούν να συμμετάσχουν. Τέλος, ξέρουμε ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής και των στόχων της ε, πρωτεύουσας, όπως ε, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αίσθησης του ανήκειν, υποστήριξη ισχυρότερων δεσμών και τέλος είστε όλοι πρεσβευτές αυτού του τίτλου. Μπορείτε να πάτε στα, στις εκλογικές σας περιφέρειες, ε, να ε, κάνετε μία εκστρατεία για να είναι υποψήφια η πόλη σας. Θα είχα κι άλλα να σας πω, αλλά μου πέρασαν τα 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω μέσα από τις ερωτήσεις ε, να κάνουμε τις ευρωπαϊκές πόλεις ε, πιο νεανικές μαζί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Και τώρα ξεκινάω τον γύρο των ερωτήσεων. Το ερώτημα είναι πώς εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού μπορούμε να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε στο ε, επίπεδο του προγράμματος Discovery U να δούμε όχι μόνο το θέμα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτεύουσών, αλλά και των ευρωπαϊκών ε, ε, πρωτεύουσών νεολαίας. Και μέσα από το Horizon να έχουμε περισσότερη εμπλοκή των νέων σε δραστηριότητες, να κάνουμε ταξίδια προς τις πόλεις αυτές να υπάρχει μια τακτική ανταλλαγή με τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Νεολαίας ε, όπως μας παρουσιάσατε εδώ στην Επιτροπή μας, έτσι ώστε οι δραστηριότητές σας και τα συγκεκριμένα project ε, που προκύπτουν αυθόρμητα να μπορούν μετά να βρουν μια συνέχεια μέσα από την Επιτροπή μας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Έχω ήδη δύο ε, που ζητούν το λόγο, η κυρία Καμέβερτ, η κυρία Ζόρζαμα και κυρία Φαράν, όχι, όχι. Η συνάδελφό σα. Η κυρία Κάμερ Έβερτ και μετά η κυρία Ζόρκοβα. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και πραγματικά για τη δέσμευση ε, που έχετε επιδείξει σχετι... ως Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας ε, για το θέμα των Ευρωπαϊκών Πρωτεύουσων Νεολαίας. Τώρα για την ερώτηση πώς μπορούμε εμείς ε, να κάνουμε από κοινού πιο γνωστή την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για να έχει αντίστοιχη αξία με την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Πραγματικά, καλό θα ήταν να το σκεφτούμε. Αυτό βοηθά και για την... Ε, ε, δεν θα βοηθήσει πολύ, βέβαια, ε, την δημοσιότητα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας εγώ ήθελα να σας ρωτήσω προς το παρόν τι κάνετε για να φτάσετε στους νέους, ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιείτε, πάτε μέσα από ε, ενώσεις, συλλόγους νέων. Ε, επίσης, κατά την εμπειρία σας, πόσοι νέοι τελικά κάθε χρόνο πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας και λαμβάνουν μέρος της δραστηριότητας, για να μπορέσουν όλα να γίνουν σωστά, θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες, έτσι ώστε να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να βγει πιο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας πούμε, στην ε, Γερμανία, στην αρχή του χρόνου, αναφέρεται ποιες είναι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ίσως ε, να κινητοποιηθούμε και να πούμε ότι δεν υπάρχουν μόνο οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Νεολαίας. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι ε, και τα μέσα που τους εκπροσωπούν στην Ευρώπη θα μπορούν να κινητοποιηθούν. Απ' την άλλη, μπορούμε να πούμε ότι και εμείς στην Επιτροπή θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε και να δώσουμε όσο μεγαλύτερη δημοσιότητα γίνεται. Όσον αφορά να μπει στο Discover EU το θέμα αυτό, αυτή την πρόταση την έχουμε κάνει ήδη, θα ήταν καλύτερο όμως ως προσέγγιση να ξεκινήσουμε με μία επίσκεψη για να δούμε αν μπορεί να μπει όσο υποχρεωτικό αυτό το ταξίδι για το Discovery U. Καλό θα ήταν λοιπόν να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις σχετικά με το τι κάνετε ήδη για να μπορέσουμε μετά εμείς επιπλέον on top να βάλουμε κάποια πράγματα και να κινήσουμε, να κινητοποιήσουμε το κοινό ε, υπέρ αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας. Δεν έχω πολλές ερωτήσεις, οπότε κάνουμε ping-pong. Πρώτα μία ερώτηση, μετά μία απάντηση και ούτω καθεξής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much for the question. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και για την υποστήριξη όσον αφορά τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσα Νεολαίας. Απάντηση, βασιζόμαστε πολύ σε άλλους οργανισμούς που είναι μέλη. Είμαστε τεράστιο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε Εθνικά Συμβούλια Νέων και Διεθνείς Οργανισμούς Νέων και έχουμε τα δικά μας μέλη. Τεράστια πηγή, τεράστια πλατφόρμα που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οργανώνουμε και εκδηλώσει και σε διάφορε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε νέων. Πώ προσεγγίζουμε του νέου. Χρειαζούμε διάβλου επικοινωνία, ενθαρρύνουμε άλλου εταίρου να μοιραστούν πληροφορίε για τι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε νεολαία. Έχουμε ε, μια επιτροπή ε, για την επιλογή των πρωτεύουσών και ζητάμε από τα μέλη των διαφόρων φορέων να μας υποστηρίξουν ότι ο τρόπος να διαδώσουν το μήνυμα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεόλεας Τώρα, πόσοι νέοι συμμετέχουν στις δραστηριότητε δύσκολο να πούμε ακριβή αριθμό. Είδατε, έχουμε 10.000 συν εθελοντέ και μετά χιλιάδε και χιλιάδες νέους που συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητε. Κάποιοι από αυτούς αφορούν τη δημιουργία δυνατικότητας, τη δική τους εξέλιξη, άλλες δραστηριότητε συμμετέχουν χιλιάδες νέοι σε φεστιβάλ και παρόμοιες εκδηλώσεις. το αριθμό των δραστηριοτήτων είναι πολύ μεγάλος. Στο Νόβι στην τελευταία πρωτεύουσα Ιανουαρία το 2019, διοργανώσαμε 1.140 δραστηριότητε το χρόνο. Μερικές από τι εκδηλώσεις ήταν μεγάλη κλίμακα, προσελκύοντα νέου και από το εξωτερικό. Αν δείτε και το, τη δημοσίευσή μας, όπω όπως Μπράγα, η Θεσσαλονίκη και το Νόβι Πρέπει εκεί να υποβληθεί τελική έκθεση, να υποβάλουν τελική έκθεση. Έχουμε αύξηση και του τουρισμού από πλευρά νέων. Πολλοί νέοι, Ευρωπαίοι νέοι, πάνε και επισκέπτονται τι πρωτεύουσε. Αν πάμε στο Κασκάι, που θα είναι πρωτεύουσα, στο, ήταν πρωτεύουσα το 2018 τη νεολαία, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και χαρήκαμε που είδαμε όλου αυτού του Ευρωπαίου που επισκεπτόταν και τους νέους να επισκέπτονται τις πρωτεύουσε Μεγάλη εμπειρία να συναντούμε άλλους νέους από άλλα μέρη της Ευρώπης και να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Τώρα για τα μέσα, για τα μίδια, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις επαφές που έχουμε με τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, αλλά πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και οι πρωτεύουσε με τα εθνικά ΜΜΕ. Δεν έχουμε εμείς την ίδια πρόσβαση που έχουν αυτές. Και είναι και θέμα πόρων. Δυστυχώς, δεν είναι το καυτό θέμα η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαία. Θέλουμε να γίνει καυτό θέμα, να προσελκύει την προσοχή των ΜΜΕ. Υπάρχει πάρα, πολύ, πάρα πολλές δυνατότητες υπάρχουν. Ελπίζουμε μέσω αυξημένης υποστήριξη υποστήριξης να πλησιάσουμε τις δυνατότητες που να χρησιμοποιήσουμε. Αυτά κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ. Μιχαέλα Ζόιντροφα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είπατε σχεδόν τα πάντα όσον αφορά τις δραστηριότητες σας. Έχετε μεγάλο ανταγωνισμό από ό,τι βλέπω. Έχουμε στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, ευρωπαϊκές πόλεις αθλητισμού και οι πόλεις που θέλουν να γίνουν ευρωπαϊκή πόλη για κάποιο θέμα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες. Δεν ξέρω αν θα θυμόσαστε το Κόσιτσε στην Σλοβακία, Ευρωπαϊκή Πόλη της Νεολαίας. Και εκεί είχαν οργανωθεί μεγάλες εκδηλώσεις, σημαντικοί εορτασμοί και έδωσαν ιδιαίτερο τόνο στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, έχετε την υποστήριξή μας. Συμφωνούμε με την ιδέα της Προέδρου μας, δηλαδή ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για δικτύωση πρέπει ο ανταγωνισμός αυτός να έχει καλά αποτελέσματα. Θα δούμε τι θα δώσει το μέλλον. Αναφερθήκατε στον προϋπολογισμό στα κονδύλια που απαιτούνται για την ορατότητα. Τα χρήματα στα πλαίσια του έρασμος. Στα πλαίσια του σώματος αλληλεγγύης τη χρηματοδότηση επίσης αναφέρατε θα μπορούσαμε να έχουμε και προγράμματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού για την επίτευξη στόχων και οι νέοι θα μπορούν να συναντώνται σε αυτά τα νέα πλαίσια. Νέα προγράμματα θα μπορούσαν να δρομολογηθούν και να είναι στη διάθεση των νέων. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι ενδεχόμενα εμπόδια που θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε. Και θέλω να πω ότι μπορείτε να βασιστείτε στην Επιτροπή μας. Θα σας στηρίξουμε σαν Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Σοϊντρόβα για τις ε, ε, ερωτήσεις σας. Ο ανταγωνισμός είναι καλός γιατί μας κάνει να προσέχουμε διάφορα θέματα. Δεν θέλουμε να είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Όπως είπα και στην παρουσίασή μου, το Ρότερνταμ ξεκίνησε αυτή η ιδέα με την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Νεότητας. Προσπάθησαν εκεί ε, οι νέοι να συμμετέχουν πιο πολύ και να πάρουν τα ενία στην πρωτεύουσα που ζουν. Όσο περισσότερη σχέση έχουμε με τις πρωτεύουσες αυτές, με τις πόλεις αυτές, τόσο το καλύτερο. Αναδεικνύουμε τις διάφορες πλευρές της Ευρώπης, ε, προσεγγίζουμε τον τοπικό πληθυσμό, ενισχύουμε την αγκίστρωση ε, της ευρωπαϊκής ιδέας στον απλό πολίτη. Αναφερθήκατε στο Erasmus Plus και στα διάφορα άλλα προγράμματα. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής, πράγματι. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε δηλαδή τεχνικά ε, πώς, ποια μορφή θα λάβουν όλα αυτά με την ανακάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα οι νέοι όταν ταξιδεύουν μπορούν να περάσουν και από την Ευρωπαϊκή ε, Πρωτεύουσα Νεολαίας. Υπάρχει και το Σώμα Αλληλεγγύης. Μπορούμε να δούμε τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής, τα τεχνικά του θέματος. Το σημαντικό είναι να το στηρίξουμε, να ε, χυθεί απλέ το φως, δηλαδή τα φώτα των προβολέων σε κάθε πόλη να στραφούν προς αυτό το πρόγραμμα για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, ναι. μεγαλύτερη δημοσιότητα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά που έχουμε καταφέρει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων. Όμως, σε συνθήκες αυξημένου ανταγωνισμού. Πώς μπορούμε αυτό να το διατηρήσουμε. Έχουμε ένα άτομο πλήρους απασχόλησης. Ε, μαχόμαστε να έχουμε πρόσβαση ε, στα ΜΜΕ, δίνουμε μάχη. Πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε διαφορετική κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος δεν ε, στοχεύει στο ίδιο πράγμα η κάθε πρωτεύουσα νεολαία. Δεν είναι το ίδιο μέγεθο σε κάθε πόλη. Δεν έχει τι ίδιε ικανότητε και δυνατότητε. Την πρώτη φορά είχε δοθεί σε πρωτεύουσα, πράγματι, στα τύρανα τη Αλβανία. Ε, μετά όχι. Ε, αλλάζει δηλαδή το παιχνίδι κάθε φορά και αυτά είναι τα εμπόδια, πώς αυτό το χαρακτηρισμό, αυτό το τίτλο Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νέων μπορούμε να το δώσουμε και σε μεγαλύτερες πόλεις από τη μία χρονιά στην άλλη, να αυξήσουμε την ορατότητα αυτού του εγχειρήματος. Θέλουμε να δουλέψουμε και με εσά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με οποιονδήποτε άλλο φορέα τυχόν ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιώβεβα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ από την πλευρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Ανήκω και εγώ στη νεότερη γενιά και βεβαίως συμφωνώ με αυτό που λέτε. Πολλά μένει να γίνουν και πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν. Το είπατε κι εσείς. Από νέους για τους νέους. Συμφωνώ απολύτως με αυτή την παραδοχή. Εξού και βρίσκομαι εδώ, εξού και ασχολούμαι με την πολιτική. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, ε, υπάρχουν πιο πρακτικές, πιο συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα αποκαταστήσουμε, πώς θα καλύψουμε αυτό το κενό στην ορατότητα. Θέλουμε να απευθυνθούμε στους νέους, να φτάσουμε μέχρι σε αυτούς, να έχουμε πρόσβαση στους νέους που δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάζονται και με τους πολιτικούς, ε, ίσως να έχουμε περισσότερες επισκέψεις. Κλειδί είναι να δουλέψουμε επιτόπου στο πεδίο. Να τους φέρουμε εδώ. Να μας δουν ότι είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι που απλά θέλουμε να βοηθήσουμε. Αν τώρα η πραγματικότητα που βιώνεται καθημερινά είναι τελείως διαφορετική από τις παρουσιάσεις που ακούμε εδώ, πρέπει να μας το πείτε. Συμφωνώ με τις ιδέες που αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την νεολαία και εγώ ενίοτε δυσκολεύομαι πολύ. Νομίζω όμως ότι πρέπει να έχουμε στόχο τη δημιουργικότητα, να αλλάξουμε το γλωσσικό ιδίωμα που υιοθετούμε όταν απευθυνόμαστε στη νεολαία. Και βεβαίω μπορείτε να βασιστείτε στη στήριξή μα. Το είπαν και οι προελαλήσαντε. Συμφωνώ με αυτού. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σα απευθύνω. Οι εμπειρίε που αποκομίζετε ανά τι χώρε. ανά τι πόλεις, ανά τι χωρε πω τι μοιράζεστε, πω τι διαπεριβάζετε. Αναφέρομαι στι βέλτιστες ή στι καλέ πρακτικέ που προκύπτουν από αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Απάντηση. Η κυρία Γιονουσάιτε. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Πράγματι, χρειαζόμαστε τη στήριξη των θεσμικών οργάνων για να ενισχύσουμε την ορατότητα του προγράμματός μας. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή των Περιφερειών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις τοπικές κοινοτικές, ε, δημοτικές και περιφερειακές ε, αρχές. Βασιζόμαστε στα μέλη να διαδώσουν το μήνυμα ε, στις χώρες τους και προσπαθούμε να απευθυνθούμε στις τοπικές αρχές και να τους πούμε ότι πρέπει να έχουμε εταιρικέ σχέσεις με τους νέους και τις οργανώσεις νέων, γιατί αυτοί είναι οι δύο φορείς που πρέπει να μπουν στο τρένο, με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούμε στενά. Και τελικά, περί αυτού πρόκειται άλλωστε σε αυτόν τον ανταγωνισμό για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα, για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων. Όλα αυτά στηρίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπάρχει όντω ανταγωνισμό ποια πόλη θα πρωτοπροβληθεί, ποια πόλη θα αναδειχθεί και πρέπει εμεί να προσπαθήσουμε να αναδειχθούμε, να αναδείξουμε το πρόγραμμα το πρόγραμμά μας. Ε, είναι με πολύ καλή πρέσβηση οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυτές καθεαυτές που διαδίδουν αυτή τη γνώση, αυτό το μήνυμα και εμπνέουν. Και αυτό είναι και η απάντηση στο ερώτημά σα για το πόσο μοιραζόμαστε τι καλέ πρακτικέ. Υπάρχει δηλαδή ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πρωτευουσών που ενώνει τι πόλει τι οποίε έχει αποδοθεί αυτό ο χαρακτηρισμό. Και μόνο μία πόλη εδώ από αυτές που αναφέραμε διαθέτει αυτό το τίτλο, αυτό το χαρακτηρισμό κάποια άλλη θα έχει την ευκαιρία να το υλοποιήσει στο μέλλον. Άρα οι πόλεις αυτές δημιουργούν ένα δίκτυο και δουλεύουν με βάση project, με βάση συγκεκριμένα έργα. Μοιραζόμαστε μέσω αυτού του δικτύου της εμπειρίας και ε, έχουμε την ε, διανοητική παραγωγή που προέκυψε μετά από αυτή τη θητεία της εκάστοτε πόλης με την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας. Και έτσι μοιράζεται αυτή η γνώση και διαδίδεται. Οι πόλεις δηλαδή είναι οι καλύτεροι πρέσβεις για να εμπνεύσουν και οι νέοι βεβαίως. Ακούσαμε πολλές ιστορίες και βλέπουμε και τις αιτήσει Και μας λέει, γράφει ένας νέος, ότι πήγα σε αυτή την εκδήλωση και έμαθα, συνάντησα ένα νέο που είναι από τυχή Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα και μου μίλησε για το project που κάνουν, για αυτές τις δραστηριότητες και με ενέπνευσε, με ενθουσίασε και γι' αυτό εγώ τώρα ορμόμενος από αυτό το περιστατικό θέλω να υποβάλω τη χύψη αίτηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και είναι πολύ καλά. Ο κύριος Μπαλάτε. Κοιτάξτε, όντω χρειάζεται στήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γραφεία σύνδεση σε κάθε χώρα μέλο και μπορεί να διαδώσει αυτό το μήνυμα, να μεταφράσει το μήνυμα στη, στη γλώσσα της χώρας ε, και ε, να ε, αναπτύξει δράσεις με τους τοπικούς φορείς. Και αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα, όπως μου ζητήσατε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γενμπού. Και εγώ σας ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Είχα την ευκαιρία να πάω στην Αμιένη στις 26 Ιανουαρίου μετά από πρόσκληση δική σας για το φόρουμ. Και μπόρεσα έτσι να δω τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται. Υπήρχαν εργαστήρια. Οι νέοι είχαν δουλέψει πάνω σε προτάσεις. πολιτισμός, εκπαίδευση και κοινωνικά εργαλεία π.χ ήταν ένα εργαστήριο. Ο, ο συνάδελφος ο κ. Μπιτό ε, συμμετείχε σε ένα εργαστήριο για την αηφορία. Δουλέψαμε σε κύκλο. Ε, καθίσαμε κυκλικά, μας παρουσίασαν τις προτάσεις τους και εμείς κομίσαμε λίγο το ευρωπαϊκό όραμα αλλά και την ευρωπαϊκή οπτική γωνία. Είπαμε τι μπορεί να είναι εφικτό και τι ίσως δεν ήταν και τόσο πολύ εφικτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Γαλλία. Ήταν εξαιρετικά θετική έκθεση, πάρα πολλά εργαστήρια, πάρα πολλοί συμμετέχοντες, δεν υπήρχε θέση για όλους. Στη συνέχεια το feedback ε, που λάβαμε ήταν εξαιρετικά θετικό για όλες τις εργασίες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ε, ε, ημέρας. Εγώ δέχτηκα προσωπικά άπειρες ευχαριστίες από νέους οι οποίοι ενθουσιάστηκαν που μπόρεσαν να δουν από κοντά ευρωβουλευτή. Δηλαδή η ορατότητα έτσι ενισχύεται. Πρέπει ο βουλευτής να μετακινείται, να ταξιδεύει, να πηγαίνει στον κόσμο να τον συναντά. Έχουμε ε, και εμείς το ρόλο να διαδραματίσουμε, να μετακινηθούμε συλλογικά ή και ατομικά, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Κάτι το αρνητικό τώρα θα ήθελα να θίξω. Τους ίδιους νέους βλέπουμε πάντοτε σε αυτές τις εκδηλώσεις για τον νέον. Δηλαδή, είναι αόρατοι οι νέοι του οποίου αφορά, αλλά οι οποίοι έχουν άλλα πράγματα να κάνουν ε, δυστυχώς ε, και αυτούς δεν τους βλέπουμε ποτέ, είναι αόρατοι. Πώς θα φτάσουμε δηλαδή στους νέους που είναι πιο απομακρυσμένοι, που είναι από ε, κοινωνικές ομάδες ευπαθείς, από ε, μειονεκ... περιοχές που μειονεκτούν δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται, σημαίνει ότι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση και δεν έχουν και τη δυνατότητα. Θυμάμαι ότι στα τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια η ύπαρξη του Εράσμους ε, δεν ε, είναι ορατή, δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται, ε, δεν, δεν έχουν τέτοια στοιχεία, δεν έχουν τέτοιες πληροφορίες και πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά, να ψάξουμε, να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους από τα τεχνικά, τα επαγγελματικά λύκεια, τον οποίο ο λόγος είναι σημαντικός και πρέπει να ακουστεί σε επίπεδο κοινωνίας. Δεν ξέρω αν τους έχετε εντοπίσει, αν έχετε κάποιες ιδέες για το ποια θα ήταν η λύση, πώς μπορούμε να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς μπορούμε να βρούμε αυτούς τους νέους, να τους εμπλέξουμε επιλέξουμε στο εγχείρημά μας, ίσως ε, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ίσως με τις τοπικές αρχές, για να μπορέσουν και να μετακινηθούν. Δηλαδή είναι μια ερώτηση επί της ουσίας αυτή, να μην βλέπουμε συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους που έχουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Um, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Θα ξεκινούσα εγώ αναφέροντας το εξής. Οι διάφορε πρωτεύουσε νεολαίε τη Ευρώπη ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση τα προγράμματά του και έχουμε υπέροχα παραδείγματα. Όταν εστιάζονται οι πρωτεύουσε επί των νέων που συνήθω δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, που δεν είναι ενεργοί στην κοινωνία. Το Κασκάι, κατά την άποψή μου, είναι πραγματικά ένα πολύ καλό παράδειγμα. Εστιαστήκαμε επί γεφυρώματος του χάσματο μεταξύ των νέων που ζουν στο κέντρο τη πόλη και εκείνων που ζουν εκτός στην περιοχή του Κερκεβέλος. Δεν ξέρω αν προφέρω σωστά την περιοχή, στα πορτογαλικά. Όταν πήγα εκεί, έκανα αυτό που κάνουμε σαν φόρουμ της νεολαίας. Πάμε σε αυτές τις πόλεις να, κάνουμε, να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις, να συναντήσουμε τους νέους, να δούμε πώς τα πάει η πρωτοβουλία μας, τι αντίκτυπο έχει στη ζωή τους η πρωτοβουλία μας. Και είχα την τιμή να πάω και να μιλήσω με αυτούς τους νέους. Συνάντησα νέους που έγιναν ενεργοί λόγω της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας νεολαία διότι η πόλη επένδυσε πολλά για να προωθήσει το γεγονός. Στην εκδήλωση χρησιμοποίησαμε κοινωνικούς λειτουργούς, κέντρα νέων και πραγματικά πλησιάσαμε τους νέους εκτός της, ε, του κέντρου της πόλης προτείνοντάς τους δραστηριότητες που μας ενδιέφεραν. Ήθελα αυτό να μοιραστώ το υπέροχο παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά στο Κασκάις προσπαθήσαμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, εκεί εστιαστήκαμε. Τι κάνει το European Youth Forum. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία. Όταν υποβάλλονται αιτήσει, έχουμε διάφορα βήματα. Κάνουν αίτηση οι πόλεις και ανάλογα με την άποψη των, της Επιτροπής και των ειδικών Προσπαθούμε να βελτιώσουμε διάφορε πτυχέ να προτείνουμε. Θέλουμε το πρόγραμμα να έχει συμπεριληπτικό χαρακτήρα, να πλησιάσουμε του νέου. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τι πόλει να αναπτύξουν κατάλληλα προγράμματα και δραστηριότητε. Πραγματικά πλησιάζουν περισσότερου νέου που κανονικά δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Διότι θεωρούμε ότι ο τίτλο αυτό Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαία αφορά όλου του νέου όχι μόνο στην πόλη, αλλά στην περιοχή, στην περιφέρεια, στη χώρα, στην Ευρώπη. Αυτό κάνουμε, δημιουργούμε τη δυνατότητα στις πόλεις να κατανοήσουν οι πόλεις τι εργαλεία μέσα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πλησιάσουν περισσότερους νέους. Σαν το Φόρουμ Νεολαίας, δεν έχουμε την απάντηση την αποκλειστική, δεν έχουμε μία μοναδική λύση, δεν έχουμε την ασημένια σφαίρα. Ε, θα παίρναμε το βραβείο Νόμπελ αν βρίσκαμε τη μοναδική απάντηση, αλλά προσπαθούμε διάφορα πράγματα και αυτό είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους κινούμαστε. Πράγματι, ζητάμε από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσε νεολαίας να εστιάζονται επί διαφόρων ομάδων, όπως είπατε, ε, διάφορα επαγγελματικά ε, λύκεια και άτυπες ε, προσεγγίσεις. Να πλησιάσουμε τους νέους που δεν είναι πραγματικά επίσημα δραστηριοποιημένοι σε σχολεία και λύκεια επαγγελματικά κλπ και είναι ένα εργοτάξιο. Πάντα έχουμε εξελίξεις, πάντα προχωρούν τα πράγματα και αλλάζουν. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να, να απαντήσω στην άλλη ερώτηση, λοιπόν, της κ. για τη συμπερίληψη. Είναι μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο πρόβλημα. Η στόχη η μελλοντική του Erasmus Plus. Να επενθυμίσω ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της, πρόταση κανονισμού για το Erasmus Plus μετά το 2020 ε, έδειχνε ότι ο καλύτερο τρόπο να προσεγγίσουμε του πλέον ευάλωτου νέου ήταν οι χώροι που ενθαρρύνουν την ε, άτυπη εκπαίδευση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή όλοι μαζί τις παραμονές έκτακτου Συμβουλίου Ευρωπαϊκού για να επενθυμίσουμε ότι χρειάζεται παραπάνω πόρου στο πρόγραμμα Erasmus για να καλύψει αυτή την ανάγκη, αυτή την πρόκληση. Να μην λησμονούμε ότι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες νεολαίας εμείς δεν δούμε τεράστιους όγκους πακτολούς χρημάτων για να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα. Γίνονται επενδύσεις των Δήμων και των πόλεων. Από την τσέπη τους πληρώνουν. 7 εκατομμύρια ευρώ για ένα χρόνο, παραγματος χάρη, σας λέω, σαν παράδειγμα. Υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες πόλεων και εργασιών. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό. Η υποστήριξη στις οργανώσεις νέων, τις επιτόπιες, τους συνδέσμους, κατάρτισης κλπ. Η επαφή μαζί τους μας βοηθά να προχωρήσουμε πιο πέρα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό πάντα από όταν εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ γίνονται διάφοροι με τις φορές νεολαίες προσπάθειες να προσελκύσουμε τους νέους οι οποίοι είναι σε δυσμενή θέση προσπαθούμε να τους δώσουμε θέση στα κέντρα αποφάσεων όσον αφορά την ορατότητα. Θέλατε να είμαστε πρέσβεις της προσπάθειας που γίνεται να πηγαίνουν επιτόπου εδώ και τρία χρόνια σε κάθε άνοιγμα, τελετή έναρξης της πρωτεύουσα, πάντα ένας ε, επικεφαλής κυβέρνησης, πρωθυπουργός, ελάμβανε το λόγο, έκανε ομιλία. Το κάναμε στην Πορτογαλία, στη Σερβία, στη Γαλλία, στην Αμιένη πες. Δεν μπορούμε να σας εθαρρύνουμε να γίνεται αυτό. Και τους συναδέλφους και τους παρόντες και τους άλλους ε, να γίνεται αυτό και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζόιτχοβα. Δεν έχω ερωτήσεις. Να διορθώσω ένα λάθος που έκανα. Ανέφερα το Κόσιτσε σαν Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Το Κόζιτσε στην Ανατολική Σλοβακία είναι Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Εθελοντισμού για το 2019. Βέβαια, εθελοντισμός και νεολαία είναι πολύ κοντά και μπερδεύτηκα. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας και ε, καλή τύχη στις προσπάθειές σας. Η κυρία Σεμέντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την παρουσίαση. Να πω, ως πρώην ε, δημοσιογράφος της τηλεόρασης, πραγματικά το να βλέπεις ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση στα ΜΜΕ και όταν ε, υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή στα εργαστήρια είναι πραγματικά σημαντικό. Θα ήταν μια ιδέα να το κάναμε αυτό. Το είπατε ήδη, οι νέοι πολιτικοί να εμπλακούν. Ίσως να υπάρχει μια εβδομάδα focus ή τρεις μέρες, ε, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτή την πόλη βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Νεολαία. Αυτά μόνο για τα ΜΜΕ. Έτσι σαν ε, συμβουλή το δίνω. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει ήδη σχεδιαστεί ή όχι κάτι τέτοιο. Ε, λίγο με απογοητεύει που το Λουξεμβούργο δεν είναι εκεί στον κατάλογο, αλλά ήδη η, Πορτογουλ... η Πορτογαλία έχει γίνει δύο φορές ε, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Δύο πόλεις. Ε, πραγματικά θα ήθελα να μάθω οι οργανώσεις νεολαίας στην Πορτογαλία ή τέλος πάντων οι τοπικές κοινότητες τι κάνουν διαφορετικό για να μπορέσουν δύο φορές να οργανώσουν ε, τέτοια ε, δραστηριότητα και να υποστηρίξουν τους νέους στην Ευρώπη. ο, θα, ο συνάδελφος θα ξεκινήσει. Όσον αφορά την ορατότητα, το να είναι όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί αναφέρθηκε και στην παρουσίαση πηγαίνουμε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πρωτεύουσες της νεολαίας, ε, πάνω από 200 νέοι ε, κάθε φορά, μία φορά το χρόνο και μιλάμε για διάφορα πράγματα. Και προσκαλούμε και τα ΜΜΕ, αλλά για κάποιο λόγο δεν βλέπουν την πρόκληση. Πραγματικά, αν μπορούσατε να μας δώσετε τα κολπάκια και τις συμβουλές που θα μας βοηθούσαν να τους προσελκύσουμε, ε, θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε μετά τη συνεδρίαση. Τώρα για την Πορτογαλία, ναι όντως είχαμε δύο πόλεις από την ίδια χώρα και αν είδατε τον κατάλογο έχουμε και τη Ρουμανία και άλλη μια που έχει γίνει μια φορά ήδη πρωτεύουσα και άλλη μια πόλη από τη Ρουμανία που έχει ζητήσει, υποψη... έχει θέσει υποψηφιότητα τι γίνεται ε, κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. Έχουμε τους ε, νέους που συνεργάζονται με τους πολιτικούς ενεργά. Αυτά είναι μια καλή διάσταση. Ε, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το Youth Work Youth Policy σχετικά νωρίς και η Πορτογαλία είναι μια από τις πόλεις που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των νέων πολύ. Είναι κομμάτι της νοοτροπία τους ότι οι νέοι και οι πολιτικοί πρέπει να συνεργάζονται. επίση στην Πορτογαλία είναι ας πούμε το μοτίβο ε, κατά κάποιο τρόπο οι νέοι πολιτικοί να προέρχονται από τις τάξεις των οργανώσεων των νεολαίων ε, από τις τοπικές κοινωνίες και να μπαίνουν στον πολιτικό στίβο. Νομίζω ε, στο Κασκάις, για παράδειγμα, το τμήμα της νεολαίας είναι το μεγαλύτερο στη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30 άτομα που δουλεύουν εκεί. Αλλά δεν έχουν πολύ δήμοι το ίδιο. Το ίδιο και στην Πράγκα. Η Μπράγκα είναι πραγματικά πρωταθλήτρια για τους νέους στη χώρα σε επίπεδο δηλαδή δραστηριοτήτων και project, αλλά και στο επίπεδο της υποστήριξης που λαμβάνουν από τις ντόπιε αρχές. Είναι τα καλά παραδείγματα από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον που να θέλει το λόγο. Τελειώνοντας να πω ότι ε, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε και στη φάση της διαφήμισης, αλλά και εκ των υστέρων θα ήταν καλό να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους νέους ε, στις ευρωπαϊκές πόλεις, τι απομένει, ποιες ε, είναι οι δραστηριότητες ε, που λαμβάνουν χώρα ήδη και ποιες θα μπορούσαν να γίνουν. Μπορεί να πει κανείς ότι όλα έχουν φτάσει σε ένα ύψιστο επίπεδο, όμως θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες για τους νέους που θα μπορούσαν να βελτιώσουν στο διηνεκέ στην κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαία. Ε, τι θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι και πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε. Um, so it's a very Πολύ καλό το ερώτημα. Σας ευχαριστώ για αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Άλλο είναι να υποβάλει αίτηση μια πόλη και άλλα είναι αυτά τα που τους ρωτάμε όταν τους συναντούμε, τους ρωτούμε. Ποιο θα είναι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος. Γιατί αυτός ο τίτλος, αυτή η ιδιότητα είναι ένα σημείο έναρξης για να πυροδοτήσει αλλαγές σε μια πόλη και οι αλλαγές δεν συμβαίνουν μέσα σε μια, σε μια χρονιά. Είναι κίνητρο όμω για τις πρωτεύουσε και τις πόλεις να συνεχίσουν να δουλεύουν και μόλις λήξει αυτή η χρονιά. Ε, Φυσικό είναι ο αριθμός των δραστηριοτήτων να μειώνεται. Μένει όμως η σημαντική κληρονομιά, οι δομές. Σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νέων, το αναφέραμε και στην παρουσίασή μας, πρέπει οι πόλεις να χτίσουν δομές στις οποίες να συμμετάσχουν νέοι και να διαχειριστούν και να διοικήσουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σε ισότιμη βάση με, έχοντας τους εκπροσώπους των δημοτικών αρχών ως ομολόγους. Στόχος είναι να προσελκύσουν ευρωπαϊκές ενισχύσεις για δραστηριότητες της νεολαίας, για αύξηση πόρων, για δημιουργία δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Άλλοι φορείς παραμένουν περισσότερο πολιτικής απόχρωσης και εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η κληρονομιά όμως είναι σαφής, είναι πρακτική και συγκεκριμένη και τη βλέπουμε σε κάθε πόλη να υπάρχει. Εξαρτάται από τις ανάγκες δηλαδή της κάθε πόλης. Μιλήσαμε και για το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πρωτεύουσων Νέων. Συνεχίζουν τη δουλειά σε αυτό το δίκτυο και μετά που θα λήξει αυτή η θητεία. Έχουμε και το συμμετοχικό προϋπολογισμό, τη συλλογική χρηματοδότηση. Δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά μπορούν οι νέοι να το αξιοποιήσουν και να αποφασίσουν ποιο μέρο του προπολογισμού θα στραφεί προς ποιες δραστηριότητες, ποιε είναι αυτές που θα υλοποιηθούν. Οι ίδιοι θα κληθούν να τι υλοποιήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή η κατά σε γενικές γραμμές είναι η κληρονομιά. Θέλουμε χώρους για τους νέους με βάση τις ανάγκες τους. Οι νέοι συνεργάζονται υπάρχουν στις πόλεις και συχνά τους λείπει χώρος. χώρος. Στο Τωρίνο ήταν η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων το 2010 και τα κέντρα νεότητας υπάρχουν ακόμα και σήμερα και τα διαχειρίζονται νέοι. Ε, εξαρτάται και από τις γνώσεις. Αλλά οι νέοι αποκτούν δεξιότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γίνονται ακτιβιστές, μπαίνουν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας, μπαίνουν πιο εύκολα στην πολιτική. Συμβαίνει αυτό και στην Πορτογαλία και αλλού σίγουρα είναι πρόκληση. Γιατί μειώνεται η διαθέσιμη χρηματοδότηση μετά το τέλος της χρονιάς. Θέλουμε όμως να έχουμε μια βάση, τα θεμέλια για να ξεκινήσει κανείς και ελπίζουμε ότι αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, θα είναι κίνητρο να συνεχιστούν οι δραστηριότητες και μετά τη λήξη του έτους. Ευχαριστώ. Στο τέλος η κυρία Φλωρένσια Φανχάουτα από την πλευρά της Επιτροπής και το ίδιο ο κύριος ε, Στέφαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας για την όλη συζήτηση. Μεγάλο παράδειγμα του πώς μπορούν να γίνουν βάσει μιας πολύ καλής ισχυρής ιδέας και πώς την υποστηρίζουν ήδη. Πράγματι είναι μια καλή ιδέα να βελτιωθεί ορατότητα για αυτά που ήδη έγιναν και χαιρόμαστε και εμείς που θα μπορούσαμε ίσως να συμβάλλουμε και να αυξήσουμε, πιο, να βάλουμε πιο ψηλά τον πύχη. Αναφερθήκατε στη διευκόλυνση της δικτύωσης και εμείς μπορούμε να είμαστε σε επαφή με τις τοπικές ενώσεις και φορείς των νέων, να δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί, να δούμε πώς μπορούμε να εξετάσουμε τις δυνατότητες για δραστηριότητε για τους νέους αυτές τις πρωτεύουσε, όπου μπορούμε να τους προσελκύσουμε, να προσελκύσουμε νέους ταξιδιώτες να επισκεφθούν. Θέλουμε να έχουμε μια δυνατότητα να βοηθήσουμε νέους που ταξιδεύουν, να συναντήσουν άλλους νέους σε μια πόλη, ε, να συναντηθούν και να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητε που ίσως να θεωρήσουν ότι είναι ενδιαφέρουσες οι οργανώσεις των νέων τα, τα προγράμματά μας και στην πολιτική μας για την νεολαία. Ήδη προωθούμε το να πλησιάσει η Ευρώπη τους νέους σε τοπικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα Erasmus Plus υπάρχει συνεργασία όσον αφορά το ότι η Ευρώπη κινείται σε τοπικό επίπεδο. Προωθούνται προγράμματα σχετικά και υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας να προωθήσουμε το τι, να εξηγήσουμε το τι είναι η συμμετοχή των νέων και πώ μπορούν να συμμετάσχουν οι νέοι στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα μέχρι και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στο μέλλον θέλουμε να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε αυτή τη διάσταση. Ποια είναι μία από τι ιδέε μα, Να προτείνουμε προγράμματα για τη συμμετοχή των νέων και σε άλλη μορφή στο σώμα αλληλεγγύη, τα διάφορα προγράμματα αλληλεγγύη. Διότι όλα αυτά, κατά την άποψή μα, χρηματοδοτούνται με μικρά ποσά που μπορούν οι, να εστερνιστούν και να προωθήσουν και σε τοπικό επίπεδο οι ευρωπαϊκέ ιδέε. Σε κάποιο βαθμό αυτό προσπαθούν να πετύχουν και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσε ε, νεολαίας. Προσπαθούμε να εκφράσουμε μεγαλόφωνα σκέψεις και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ κύριε και γενικά ε, όλη την ομάδα σας ε, για την ε, δραστηριοποίηση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να δραστηριοποιήσετε υπέρ των νέων. Χαίρομαι πολύ για τη συνεργασία. Ελπίζω να έχουμε και άλλη συνεργασία, όχι μόνο στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας αλλά και σε άλλα προγράμματα. Ευχαριστώ. Σταματάμε λιγάκι και μέχρι να έρθει η Επίτροπος νομίζω και εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε και να κλείσουμε και τις συζητήσεις μας. Για να ξεκινήσουμε γιατί έχει φτάσει ήδη η Επίτροπος. Και όποιος δεν θέλει να μείνει, παρακαλώ να βγει από την αίθουσα. Όσοι θέλουν να συνεχίζουν τις κουβεντούλες. Να μπορούμε να έχουμε αμέριστη την προσοχή σας παρακαλώ ε, στον διαρθρωμένο διάλογο με την ε, Μαρία Γκάμπριελ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι χαρά μου που καλωσορίζω για πρώτη φορά επισήμως με τη νέα της ιδιότητα την Επίτροπο Μαρία Γκάμπριελ στο διαρθρωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πολιτικές προτεραιότητες. Έχουμε μια τακτική ανταλλαγή απόψεων μέσω των συντονιστών με τη Μαρία Γκάμπριελ εδώ και κάποιο διάστημα, όμως η επίσημη ανταλλαγή ξεκινά σήμερα και γι' αυτό χαίρομαι που είναι μαζί μας. Ε, σας καλωσορίζω λοιπόν εγκαρδίως και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην επεξεργασία του χαρτοφυλακίου σας και ειδικά στη συνεργασία με την Επιτροπή μας. Και νομίζω ότι το χαρτοφυλάκιο που σας έχει δώσει η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Φόντερ Λάιν, ε, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ε, δραστηριοτήτων. Μπορούμε να φτιάξουμε γέφυρες ε, στον επίπεδο του πολιτισμού. Βλέπω ότι έχετε ένα ε, κομμάτι. Η Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Επιτροπής, έχει βάλει τον πολιτισμό ε, μπροστά. Έχει μεγάλη σημασία. Ενισχύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ο τομέας ε, της δημιουργίας είναι αυτός ο οποίος οδηγεί στην καινοτομία, τις νέες ιδέες, έτσι λοιπόν, με μεγάλη αδημονία περιμένουμε τις ε, απόψεις σας, ε, τις δράσεις σας. Σας δίνω το λόγο για να κάνετε μια εισαγωγή και μετά θα ξεκινήσουν ερωταπαντήσεις υπό τη μορφή ping-pong. Ε, έτσι ζητώ να ξεκινήσετε λίγο με τις πρόσφατες εξελίξεις στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήταν καλό λοιπόν να ακούσουμε τι ακριβώς πιστεύει η Κομισιόν σχετικά με την πρόταση του κυρίου Μισελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ σήμερα, όπως το υπενθύμησε και η πρόεδρό σας, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την ιδιότητά μου της Επιτρόπου Αρμοδίας για την έρευνα, την ε, εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την νεολαία μεταξύ άλλων. Χαίρομαι με αυτή την προοπτική να συνεργάζομαι στενά μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου στη θέση της Επιτρόπου. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ευρώπη έχει θέσει νέους στόχους πολύ πιο φιλόδοξους στην πολιτική της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Και για να τους πετύχουμε αυτούς πρέπει να ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε ένα ανώτερο επίπεδο. Για να γίνει αυτό πρέπει να αποκτήσουμε και τα κατάλληλα μέσα για να αναπτυχθεί η συνεργασία στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να επιτευχθούν οι ανώτεροι αυτοί οι στόχοι. Θέλω να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σαφή θέση, την τεκμηριωμένη με επιχειρήματα που υιοθέτησε και για το όραμα που υπερασπίζεται έτσι ώστε η Ευρώπη να συνεχίσει να διαθέτει τα μέσα που θα της επιτρέψουν να διαδραματίζει το ρόλο κλειδί που της αναλογεί. Επιτρέψτε μου τώρα να ξεκινήσω θίγοντας ορισμένα ζητήματα, ορισμένα θέματα, προετοιμάζοντας την επίσκεψή μου σε σε εσά σήμερα, ε, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν 15 σημεία για τα οποία έχω να κάνω σημαντικέ ανακοινώσει και θα επανέλθω κατά τη διάρκεια τη παρουσίασή μου. Αλλά θέλω πρώτα να θίξω του βασικού ακρογωνιαίου λήθου. Πρώτον, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευση. Έχει προβλεφθεί να δημιουργηθεί από σήμερα μέχρι και το 2025. Πρόθεση δική μου και τη ομάδα μου είναι να παρουσιάσουμε ανακοίνωση ανακοινωθέν το Σεπτέμβριο ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνω έκκληση ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει ενεργά, θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση. Οι ιδέε σα είναι πολύτιμέ για εμά και θα τι λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Θέλουμε να άρουμε τα εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία στην Ευρώπη, να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλή ποιότητα, να μπορούν οι μαθητευόμενοι να μετακινούνται πιο εύκολα μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων των διαφόρων χωρών και σε βάθο χρόνου να αλλάξει και η κουλτούρα, το πνεύμα που διέπει την εκπαίδευση και να υιοθετήσουν όλοι αυτή την πολύ βασική αρχή της διαβίου μάθησης. Και γι' αυτό θα παρουσιάσουμε σχετική ανακοίνωση το Σεπτέμβριο, θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για νέες δράσεις και θα θέλαμε Επίση, να παρουσιάσουμε ένα νέο πλαίσιο συνεργασία με τα κράτη-μέλη σε θέματα εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Όπω γνωρίζετε, το ET 2020, το εφιστάμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο, λύγει η ισχύ του φέτο στα τέλη τη χρονιά. Πέρα από τον Ευρωπαϊκό Χώρο εκπαίδευση. πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει νέα ανακοίνωση τον Ιούνιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτέ οι δύο δουλειέ, αυτά τα δύο έργα να συμβαδίζουν, να κινούνται πάρα παράλληλα για να μην ανακαλύψουμε εκ των υστέρων ότι υπάρχουν ασυνέπειες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θέλουμε ένα πλαίσιο πολύ πιο συνεκτικό και πολύ πιο αποτελεσματικό. Στο πλαίσιο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Χώρου για την Εκπαίδευση προφανώς τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θα αναλάβουν τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία αυτή για να βάλουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Όλοι γνωρίζουμε ε, τι εστί τρίτο βάθμια εκπαίδευση, πόσο δύσκολο είναι οι νέοι μας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες υψηλού επίπεδου για να μπορέσουν να επιδείξουν αριστεία στον τομέα των σπουδών τους. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να βρουν θέση νέοι στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας η οποία αλλάζει ακατάπαυστα και δραματικά πραγματικά. Μιλούμε για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση υψηλή ποιότητα, η οποία είναι απαραίτητη για να σταθούμε στο ύψο των προκλήσεων, για να μπορούν να έχουν οι νέοι τι απαραίτητε δεξιότητε ω πολίτε και να σφυριλατήσουν πιο συνεκτικέ, πιο ενωμένε κοινωνίε. Γίνεται λοιπόν δουλειά και έχει γίνει δουλειά, αλλά παραμένει πρόκληση σε επίπεδο εκπαιδευτικό, σχολική εκπαίδευση για να υπάρξει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και επόμενο στάδιο είναι η επιδίωξή μα να βελτιωθούν τα αποτελέσματα τα σχολικά αποτελέσματα. Και πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις εξή τρει προκλήσεις. Πρώτον, να δώσουμε σε όλου τους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις βασικές τους δεξιότητες, να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς το βασικό δίπλωμα και να ενισχύσουμε την ευημερία, την καλή διαφίωση, το ευζήν δηλαδή στο σχολικό περιβάλλον. Και έχουμε μια βασική πρωτοβουλία έτσι ώστε κάθε μαθητής να αποκτήσει κάποιες, ε, ένα συγκεκριμένο επίπεδο δεξιοτήτων στις βασικές γνώσεις και επιμένω σε αυτό γιατί για τη δημιουργικότητα και για το ψηφιακό κόσμο έχουμε άλλες πρωτοβουλίες. Μιλούμε για τις βασικές γνώσεις και βασικές δεξιότητες να έχουμε μια εγγύηση για βασική εκπαίδευση. Η προσωπική μου επιθυμία είναι να αποφύγουμε τον όρο εγγύηση, γιατί έχουμε το εργαλείο εγγύηση για την νεολαία. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Θα ήθελα να πούμε ότι στο δεύτερο εξάμεινο το 2020 θέλουμε να ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό και οι ιδέε σα είναι ευπρόσδεκτε πραγματικά και για τον Ευρωπαϊκό Χώρο εκπαίδευση, όπω όλοι γνωρίζουμε πρέπει να είναι ένας χώρος καινοτόμο και συμπεριληπτικός και θα είναι μόνο άμα έχουμε εκπαιδευτικούς με πάθος, με υψηλά προσόντα, με υψηλά κίνητρα και γι' αυτό θέλω να συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη και με εσάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τους εκπαιδευτικούς και με τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε την Ακαδημία Δασκάλων και Καθηγητών, Ακαδημία Εκπαιδευτικών, το Teachers Academy. Θα είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερω και ε, ε, θα επανέλθω σε αυτό. Θέλω όσο και περισσό, όλο και περισσότερο εκπαιδευτικοί να ε, μεταφέρουν αυτή τη σκητάλη και να υψώνουν αυτή τη δάδα ελπίδας που είναι ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης. Έρχομαι τώρα στο ψηφιακό κομμάτι, στη ψηφιακή εκπαίδευση. Γνωρίζετε ότι έχω δεσμευθεί να ενημερώσω το υφιστάμενο σχέδιο δράσης, να το επικυριοποιήσω κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας μου. Καλά νέα είναι ότι θα το έχουμε ολοκληρώσει πριν τον Ιούνιο. Με την ομάδα μου έχουμε ξεκινήσει ήδη της εργασίας και η ιδέα μου είναι εξή, να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες που αποδείχθηκαν επιτυχημένες και αναφέρομαι παραθετικά στο Safer Internet for EU, το European Code Week. Ε, χρειαζόμαστε όμως και άλλες δράσεις όχι μόνο για το ασφαλές διαδίκτυο και για την συγγραφή κώδικα. Πρέπει να ε, έχουμε και άλλες ιδέες και θέλω τη γνώμη σας και τις προτάσεις σας. Ε, σε ό,τι με αφορά μια πρωτοβουλία που με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως είναι το, η τεχνητή νοημοσύνη για τα κορίτσια. AI for girls. Υπάρχει σχέδιο για τη τεχνητή νοημοσύνη. Γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπαράγει στερεότυπα και μεροληπτικά οπτική θεώρηση της πραγματικότητας, πιστεύω ότι η θέση των γυναικών σε αυτό το τομέα και των κοριτσιών είναι εξαιρετικά σημαντική. Δύο λόγια το, για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ίδρυμα Καινοτομία και Τεχνολογία. Γνωρίζουμε πόσο έχουν προχωρήσει οι εργασίε εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Θέλω να σα ευχαριστήσω για τι πρώτε θετικέ αντιδράσει σα. Σήμερα έχουμε μπροστά μα μια νέα πρόκληση. Πρώτον, να αποκαταστήσουμε κάποια σφάλματα στο Ινστιτούτο, να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερο άνοιγμα και δεύτερον να ε, μεριμνήσουμε ώστε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία και την Τεχνολογία να έχει συνέργειες με αρμόδιους όμορους γειτονικούς φορείς. Να δοθεί έναυσμα στη βιομηχανία του πολιτισμού, του θεάματος. Να υπάρξει συνέργεια με το δεύτερο πυλώνα του ορίζοντα για την Ευρώπη και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας θα πρέπει να είναι σε πλήρη ε, συνέργεια με ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Καινοτομία. Δηλαδή, εκεί που ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά υψηλός, θα πρέπει να υπάρξει δημόσια επένδυση για να ξεκινήσουν οι start και να μπορέσουν να ε, τολμήσουν. Αξίζει αυτή η δουλειά για να ευρεθεί πιο εύκολη χρηματοδότηση και να μπορέσουν όλοι να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Τώρα, δύο λόγια για τους νέους. Κάτι πολύ σημαντικό για εμένα και το λέω διότι έχουμε μια νέα στρατηγική για τη νεολαία από το 2019 μέχρι το 2027. Τι θέλουμε να κάνουμε φέτος. Θέλουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της μελέτης για την κινητικότητα των νέων που κάνουν εθελοντισμό και με αυτή τη μελέτη θέλουμε να ταυτοποιήσουμε, να εντοπίσουμε τα εμπόδια προς την κινητικότητα και την επίδειξη διασυνοριακής αλληλεγγύης και γι' αυτό έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό και θα ξεκινήσουμε δημόσια διαβούλευση για να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις. Θέλουμε να έχουμε σύσταση από το Συμβούλιο για να προτείνουμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ε, χρονιάς ένα νέο πολιτικό πλαίσιο που θα διέπει τη διασυνοριακή αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό και θα συμπεριλαμβάνει και τις περιόδους μαθητείας και την απασχόληση. Υπάρχει και ο συντονιστής για τους νέους, Youth Coordinator, και θέλω να σας πω ότι δουλεύουμε με τους υποψηφίους έτσι ώστε να έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιον στον οποίο θα αποτελέσει και το πρόσωπο και την εικόνα και το σημείο αναφοράς. Ένα τηλέφωνο δηλαδή, τον οποίο να μπορούν να καλέσουν οι νέοι και να απευθυνθούν σε αυτόν. Να αναφερθώ και σε κάποια επικουρικά θέματα. Η άθληση δεν είναι στον τίτλο του χαρτοφυλακίου μου, αλλά ξεκαθάρισα ότι θέλω να συνεχίσει η δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η άθληση, ο αθλητισμός έχει τεράστιες δυνατότητες, μπορεί να βελτιώσει την υγεία, αλλά ξεπερνά και τα σύνορα, τα σύνορα τα γεωγραφικά, τα σύνορα τα γλωσσικά, αλλά και τα διαγενειακά. Και φέτος το θέμα θα είναι η διαγενειακή διάσταση των αθλημάτων. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερες δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση, άθληση για περισσότερες και με ε, περισσότερες γενιέ, και να έχουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ της καινοτομία και της άθλησης και του αθλητισμού. Περισσότερες ιδέες για το πώς θα δοθεί συνέχεια σε αυτές τις δράσεις ή ποια είναι η σύνδεση με την πολιτιστική κληρονομιά. Καλό είναι δηλαδή να ε, κάνουμε μία κάτωψη της κατάστασης και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Θέλω να συγχαρώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους δύο συμπροέδρους για τις σχετικές πρωτοβουλίες για τον αθλητισμό. Τώρα για την ε, κουλτούρα και τον, ε, την πολιτιστική κληρονομιά. Τον πολιτισμό γενικότερα είναι ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. Έχουμε κληρονομιά, από το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχουμε μια νέα πολιτική ατζέντα για τα θέματα κουλτούρας και πολιτισμού και όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε στενά και σε βάθος. Έχουμε εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου στο Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Κληρονομιά το οποίο οργανώσαμε. Ομολογώ ότι αισθάνομαι λίγο άσχημα διότι ε, είχαμε μια συνεδρίαση τον Οκτώβριο και η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίζεται για τον Ιούνιο. Δεν φτάνει νομίζω, θα πρέπει να έχουμε πιο τακτική παρακολούθηση σε πιο συχνά χρονικά διαστήματα. Να προβληματιστούμε όμω όλοι μαζί για το ποιε δράσει πρέπει να αναλυφθούν και να παρακολουθηθούν. Αυτή τη στιγμή ξεκινούμε το νέο μα πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Κληρονομιά σε Δράση ε, μάθηση από ομολόγους σε επίπεδο περιφερειακό για την πολιτιστική κληρονομιά. Ένα άλλο θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερος και με συγκινεί και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζω να σας εφιστώ την προσοχή στην ατομική κινητικότητα και στο εργαλείο για τους καλλιτέχνες είναι πολύ ενθαρρυντικό πιλωτικό πρόγραμμα που τρέχει τα τελευταία δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τέτοιο μηχανισμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και δύο λόγια για να σας καθησυχάσω για τη στήριξη στον κλάδο ε, της μουσικής. Έχουμε την πρωτοβουλία Music for Europe, μουσική για την Ευρώπη, η οποία θα συνεχιστεί και δεν θα διακοπεί. Περιμένουμε και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε η κουλτούρα που είναι ε, το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν και ανθίζουν οι κοινέ μας αξίες ε, να μπορέσει να καλλιεργηθεί και να προστατευθεί. Τρία τελευταία σημεία είναι τα εξή που θέλω να μοιραστώ μαζί σα. Ξέρετε ότι όλε αυτέ οι πολιτικέ έχουν τεράστιο αντίκτυπο εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω όμω να ενεργοποιήσουμε ορισμένα εργαλεία για να αποκτήσουμε ορατότητα και ε, στι τρίτε χώρε. Πιστεύω στην πολιτιστική διπλωματία. Θα μπορούσε να είναι πυλώνα τη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, κατά τη γνώμη μου. Γνωρίζω ότι τα μέσα είναι πενιχρά, γνωρίζω το φαινόμενο του κατακαιρματισμού, γνωρίζω την ανάγκη να επιλεγούν πολύ σοβαρά τα θέματα θέματα, ε, διότι δεν μπορούμε να ε, δείξουμε όλο μας τον πλούτο στις τρίτες χώρες. Όμως, έχουμε την Αφρικανική πρωτεύουσα κληρονομιάς πολιτιστικής, το Μαρακές για παράδειγμα. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα πολιτιστικής κληρονομιάς, Δηλαδή είδατε πώς ένας θεσμός δικός μας τον ε, έχουμε εξάγει στην Αφρικανική Ήπειρο. Μπορούμε να σφυριλατήσουμε δεσμούς, σχέσεις, οι οποίες μας αφορούν άμεσα, γιατί πρόκειται για σχέσεις μεταξύ ανθρωπίνων όντων προπαντός. Δύο λόγια για τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι μια περιοχή ε, και θα πρέπει σε αυτή την περιοχή να προχωρήσουμε πολύ πιο μακριά έχει, υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν μιλούμε για διαπραγμάτευση μόνο με κεφάλαια η οποία εκτείνεται σε 7 ή 8 χρόνια και στο τέλος κανείς πια δεν καταλαβαίνει τι νόημα έχουν όλα αυτά. Υπάρχει κάτι το περισσότερο. Έχουμε το πρόγραμμα Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη. Έχουμε το πρόγραμμα Erasmus+. Plus. Δύο μόνο από τους έξι συμμετέχουν. Είναι ευκαιρία να τους εμπλέξουμε, να δείξουμε στους νέους αυτή, αυτών των περιοχών, αυτή της περιοχής, ότι η κινητικότητα τους ανοίγει προοπτικές και για τη χώρα τους, για τη γειτονιά τους, για την περιφέρειά τους. Τέλος, διαπραγματεύσεις για τα μελλοντικά προγράμματα, για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, για το Erasmus Plus, αλλά και για τη Δημιουργική Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να τα συζητούμε όλα αυτά από την πλευρά μου. Ε, να δείξω ότι σέβομαι απολύτω και να τονίσω ότι σέβομαι απολύτω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερω στην επεξεργασία την τεχνική των φακέλων. Και σήμερα είμαστε στις παραμονές ενός συμβουλίου, το οποίο θα ασχοληθεί με τον προϋπολογισμό. Και αυτό βεβαίως δεν το ξεχνούμε ποτέ το θέμα του προπολογισμού. Σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να μιλούμε ενωμένοι, με μία φωνή, εμείς και εσείς. Προφανώς η πρόταση του Συμβουλίου είναι απογοητευτική, σε καμία περίπτωση δεν μας επιτρέπει να είμαστε αξιόπιστοι, όχι να πετύχουμε, αλλά ούτε καν να είμαστε αξιόπιστοι στον ισχυρισμό μας ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλους και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των νέων. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος των τριών προγραμμάτων. Με αυτή την πρόταση την απογοητευτική δεν θα είμαστε σε θέση να το πράξουμε αυτό. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από εμένα να υπάρξει μια τέτοια πρόταση η οποία δεν αντιστοιχεί στις φιλοδοξίες μας, αλλά το χειρότερο είναι ότι μας απαγορεύει, δεν μας επιτρέπει ως Ευρωπαίους να ε, ε, κάνουμε τα ελάχιστα. Όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς καινοτομία, χωρίς επένδυση στην νεολαία, στην ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, στην ε, πορεία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων εν ώψη των μελλοντικών εξελίξεων, δεν θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε καμία πρόκληση, ούτε το δημογραφικό, ούτε την ψηφιοποίηση, ούτε την ε, κλιματική αλλαγή, τα θέματα περιβάλλοντας. Χωρίς τέτοιου είδους δεξιότητες, χωρίς κουλτούρα, χωρίς πολιτισμό, καμία πρόκληση δεν θα αντιμετωπίσουμε ε, σεβόμενοι τις αξίες μας, το σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη, με καινοτομία, με βούληση για εξυγχρονισμό και για ε, πορεία προς τα εμπρός. Μακρηγόρησα λίγο κυρία Πρόεδρε, Σα ζητώ συγγνώμη, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκφράσω τις απόψει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αδειμονώ για τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις Σα Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος. Είναι τόσα πολλά τα θέματα. Έχουμε μια ε, μεγάλη βεντάλια ζητημάτων και καλό θα ήταν να ξέρουμε ακριβώς ε, τη δική σας ε, θέση. Καλό είναι να ξέρουμε τη δική σας θέση, ώστε να μπορούμε και στο Κοινοβούλιο να μιλάμε με μία φωνή σχετικά με το προϋπολογισμό. Η Ursula von der έχει ήδη χαιρετήσει τις απαιτήσει του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι έχουμε ενώπιό μας πολλή δουλειά να κάνουμε για να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι ε, δεν θέλουμε έναν αρνητικό προπολογισμό σε αυτόν τον τομέα, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα ώστε το τέλος να πριτανεύσει η λογική και να ε, λειτουργήσουμε επικοδομητικά, να υποστηρίξουμε τα προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας όπως το Erasmus Plus και να μην έχουμε τόσο μεγάλες ε, περικοπές όπως φαίνεται ότι θέλουν τα κράτη-μέλη να φέρουν τώρα. Επίσης, οι νέες πρωτοβουλίες χρειάζονται χρήματα. Και εδώ και πολλά χρόνια ε, έχουμε δει ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση, οπότε σε διαρθρωτικό επίπεδο, οπότε καλό είναι που εμείς μπορούμε από κοινού να υπερασπιστούμε μια ενίσχυση αυτών των προγραμμάτων. Όπως είπα, θα κάνουμε τη διαδικασία ping-pong. Ξεκινάμε πρώτα με τους συντονιστές και μετά οι υπόλοιποι. Πρώτα η Μιχαέλα Ζόιντροβα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, για το διάλογο μαζί σας. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε σε πολλά θέματα. Καλύψατε ευρύ πεδίο. Επιτρέψτε μου να είμαι πιο καλά εστιασμένη. Οι κανόνες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, Έρασμος, Δημιουργική Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Είναι προγράμματα πολύ σημαντικά για μας. Ο πολιτισμός, η παιδεία και η νεολαία. Πιο συγκεκριμένα, απογοητεύτηκα αρκετά. Διότι δεν συνεχίζουμε με τον ίδιο ταχύ ρυθμό που θα θέλαμε. Θέλω να πω ότι χρειάζεται επιτάχυνση. Χρειάζεται επιτάχυνση η νομοθετική διαδικασία. Για την ώρα έχουμε κάπως κολλήσει ήδη. Δεν έχουμε πετύχει συνένεση όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Δεν θα πω ότι δεν συνεχίσαμε. Αντιθέτως, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέρμα. Αλλά αυτό που απομένει είναι ο προπολογισμό, άλλο θέμα αυτό, αλλά απομένει το θέμα της διακυβέρνησης. Η ισορροπία αρμοδιοτήτων ισορροπία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Βεβαίως, σεβόμαστε τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Και θέλουμε και εμείς να συμμετάσχουμε στις ε, αρμοδιότητες επιρροής, ελέγχου. Θέλουμε να επηρεάζουμε και να ελέγχουμε κατά κάποιο τρόπο τις πολιτικές αποφάσεις. Εν ονόματι του εισηγητού και των συνεισηγητών ζητούμε μία επιτάχυνση των εργασιών. Να συμβάλλουμε στην επίτευξη συνένεσης όσον αφορά τον επιμερισμό των εξουσιών μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ο προϋπολογισμός. Έχουμε συνένεση επ' αυτού Συμφωνούμε, έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Το, η πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου, του κυρίου Μισελ, είναι απαράδεκτο. Μειώνονται τα κονδύλια. Ζήτησα λοιπόν στην επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό μας, του ζήτησα να αρνηθεί το, την πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου. Έχετε την υποστήριξή μας. Για τα νέα προγράμματα που αναφέρατε έχω μία ερώτηση. Παρακαλώ. Είχαμε πει δύο με τρία λεπτά για τις ερωτήσεις ε, αρχικά. Ε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε την ερώτηση και να έχετε και στο μυαλό σας ε, την, το χρόνο. Ε, συγγνώμη, θα κλείσω. Διότι έχουμε τον πρόεδρο διακοινοβουλευτικής ομάδας για την πολιτιστική κληρονομιά, ο συνάδελφος Μιλαμόν. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε περισσότερα για τη δράση για την πολιτιστική κληρονομιά. Θα χρησιμοποιηθεί για αποκατάσταση μνημείων, ανοικοδόμηση. Ε, μπορείτε να το διευκρίνετε, διευκρινίσετε, συγγνώμη. Και χαίρομαι για τη συνεργασία που θα έχουμε. κυρία Γκάμπριελ, ευχαριστώ για το θέμα του προϋπολογισμού. Την περασμένη εβδομάδα συνάντησα τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας Όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι οι υπουργοί οικονομικών το γνωρίζουν εδώ και τρία, τρεις μήνες το συζητώ το θέμα. Μιλώ για τον προπολογισμό του Erasmus και του Erasmus Plus και του, για το Horizon Europe. Πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ στεναροί στη θέση μας. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, ξέρετε πόσο προσπαθώ πραγματικά να βρω μια λύση. Ποιο είναι το πρόβλημα, τα τρία θέματα που μας ενδιαφέρουν, το Erasmus Plus, το Solidarity Corp και το Creative Europe, θεωρούνται σαν πακέτο μαζί με άλλα ζητήματα. Μιλάμε μαζί με άλλα εννιά. Έχουμε 12 θέματα οριζόντια. Τα συζητάμε αένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να βρούμε τεχνική αποδεκτή λύση. Και έχουμε λόγους γι' αυτό. Έχουμε επιτροπολογία, έχουμε τις εξουσίες μας, ο κάθε φορέας, πιστεύω ότι απλούστατα πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία, τη συνεργασία για να βρούμε λύση. Ξέρω ότι υπάρχει προσδοκία να κάνει πρόταση τεχνικού περιεχομένου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεχίσω να συνομιλώ με τους συναδέλφους για να βρούμε μια διέξοδο. Διότι στο κάτω-κάτω έχετε δίκιο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα βρεθούμε την 1η Πρώτου του 2021 να αντιμετωπίζουμε κίνδυνο και να λέμε δυσάρεστα πράγματα και σε αυτούς που δεν τα αξίζουν. Και το αξίζουν το λιγότερο να ακούσουν δυσάρεστα πράγματα. Βασιστείτε πάνω μου. Είναι ένα θέμα που πραγματικά είναι σημαντικό για μένα. Αλλά για μία ακόμη φορά έχουμε επιτροπολογία και κανόνε που είναι αυστηροί πρέπει να ακολουθηθούν. Πιστεύω ότι είναι δυνατό να, βούμε, να βρούμε ένα συμβιβασμό. Πρέπει να συνεχίσουμε. Από την πλευρά μου, δράτω με τη ευκαιρία να πω και να επενθυμίσω ότι όταν κάναμε προσπάθειες με τη Φιλανδική Προεδρία για να δείξουμε ότι είναι δυνατόν να προχωρήσουμε επί τεχνικών ζητημάτων, έγινε κάτι. Πρέπει να πω το ότι Discovery EU βγήκε από το Negotiating Box. Θα ήταν καλό να μπορούσαμε να προχωρήσουμε επί των τριών θεμάτων. Κατανοώ τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνδέεται με τον προπολογισμό. Για να συνοψίσω μια φράση, δεν θα πρέπει να γκρεμίσουμε τις γέφυρες, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία να βρούμε μια διέξοδο. Για το Cultural Heritage για τη σχετική δράση είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, τον Ιανουάριο του 2020 και όπως προανέφερα πραγματικά θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την εκπαίδευση του ΣΥΠΗΝ των τοπικών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω σε αυτό. Θέλουμε τις, τα quality principles να προωθηθούν να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση, τη συμμετοχική για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό που προβλέπετε για την ώρα, για το όλο πρόγραμμα, είναι να έχουμε τουλάχιστον 12 peer learning visits, επισκέψεις ομοτύπων, σε πόλεις, περιοχές επιλεγμένες στην Ευρώπη. Θα σας δώσω εγώ τον κατάλογο για να μπορέσετε κι εσείς να δείτε τι προτείνουμε. Θέλουμε να έχουμε πάνω από 20 συμμετέχοντες ανεπίσκεψη. αυτή τη στιγμή Μιλάμε για policy makers, αλλά όχι μόνο για αυτούς. Έχουμε ειδικού ε, των περιφερειών, για πολιτικές για την Ήπεθρο, rural policies, και μπορούν να κάνουν κάτι πάνω σε αυτό. Στόχος, κατάλογος με 30 καλές πρακτικές που θα μπορούσαν συνεχεία να διαδοθούν σε επίπεδο πόλεων και ευρωπαϊκών περιοχών και περιφερειών. Ξεκίνησε η προσπάθεια Δεσμεύομαι να σας δώσω τον κατάλογο αυτών των πόλεων που θα επισκεφθούμε, ποιοι θα συμμετάσχουν. Πιστεύω ότι 30 καλές πρακτικές για μένα είναι κάτι σημαντικό. Εν συνεχεία θα μπορούσα να κάνω συσχετισμούς με το Horizon Europe και τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε βάσει αυτών. Αυτή είναι η όλη ιδέα, αλλά μόλις τώρα ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος. Ευχαριστούμε. Πέτρα Καμάεβερτ. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο για πραγματικά την πολύχρωμη αυτή ανθοδέσμη ε, από θέματα που μας παρουσίασε σήμερα εδώ. Ε, ξεκινάω με το προϋπολογισμό. Έχουμε χάσει πολύ καιρό από την ε, Σύνοδο Κορυφής του ε, πριν από δυόμιση νομίζω χρόνια περίπου. Υπάρχει λοιπόν πολύ καιρός που έχουμε εισαγάγει τα θέματα για τον ορίζοντα 2020 αλλά και στην ουσία αυτό θα πρέπει να, ήδη να είχε συμβεί. Έχουμε λοιπόν ε, ε, μια σειρά από θέματα ε, τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη συγκεκριμένα στην εκπαίδευση. Έχουμε προβλήματα. Έχουμε παιδιά σε σχολική ηλικία που δεν ξέρουν ούτε να διαβάσουν. Όμως, για να μπορέσουν αυτά να τελειώσουν θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, πολύ έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα παιδιά, δηλαδή να πάρουν απολυτήριο λυκείου. Είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς απολυτήριο λυκείου, μεν, αλλά χρειαζόμαστε ε, ταυτόχρονα και χειρονάκτες. Ε, ε, πολλές φορές, λοιπόν, σε αυτά τα επαγγέλματα δεν χρειάζεται κανείς το πολιτήριο αλλά το έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να διαβάσω κάτι στο δικό σας έγγραφο. Γενικά, ε, δεν είναι καλό, θεωρώ, να λέμε στους ανθρώπους ότι μόνο όταν έχουν απολυτήριο λυκείου αξίζουν κάτι. Αυτά είναι χαζομάρες. Νομίζω επίσης, για το σημείο 3, χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για τα προγράμματα που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2021 για τη διακυβέρνηση και τα χρηματοδοτικά. Ξέρετε ότι ήδη στο Κοινοβούλιο δεν έχουμε αποφασίσει ε, οριστικά τα προγράμματα του Νοεμβρίου. Αφήνουμε για άλλη μια φορά ε, την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο να μας βάζουν εμάς μπροστά ενώ αυτοί δεν έχουν γέρος εκπληρώσει το δικό τους κομμάτι. Όχι, μα το Θεό εμείς έχουμε κάνει το δικό μας κομμάτι και περιμένουμε τις προτάσεις της Κομισιόν και τελικά παίρνουμε αυτή την απαράδεκτη πρόταση από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για το ΠΔΠ που δεν γίνεται να προχωρήσει. Πραγματικά δεν μπορούμε να μας γελιοποιείτε συνεχώς ε, κάθε φορά να έχουμε εμείς ολοκληρώσει και να μην έχετε κάνει τη δική σας, το δικό σας μερίδιο και να φτάσουμε τον Ιανουάριο και να μην υπάρχουν ε, τα χρήματα και αυτά γιατί το Συμβούλιο ε, μας έχει βάλει σε αυτή τη θέση με τις προτάσεις του για το πι δελτα πι. Πραγματικά, μα το Θεό δεν είναι δικό μας λάθος, είναι τον άλλων. Ευχαριστώ. <laughs> Merci. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο που θέσατε, για το επίγον της καταστάσεως, ένα μήνυμα που το ακούω, το καταλαβαίνω, σας ευχαριστώ να πω απλούστατα. Εάν δεν είχαμε το Αυριανό Συμβούλιο θα ήταν δύσκολο να τους ευαισθητοποιήσουμε. Ξέρουμε ποια είναι η πρόταση. Είναι απογοητευτική η πρόταση του Συμβουλίου θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Το σημαντικό που είναι για μας αυτό το πλαίσιο είναι να μην δημιουργήσουμε πανικό εκεί που υπάρχει περιθώριο λιγμών. Συνεχώς το συζητάμε με τους πρωθυπουργού, τους υπουργού, στο Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε δεν το λησμονώ. Θα συζητήσω το θέμα την ομάδα μου, αλλά από την πλευρά μου θα ήθελα αυτή την εβδομάδα να προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι σαφέ Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί πολύ και θα ήθελα πράγματι την επόμενη πενταετία να εργαστούμε περισσότερο επ' αυτού. Θα μπορούσα εδώ να αναφέρω τέσσερι πρωτοβουλίε που δεν λησμονώ, όπου εκεί η επαγγελματική κατάρτιση έχει τη θέση τη. Καταρχά, το New Skills Agenda. 25 Μαρτίου θα έχουμε το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες με τον Επίτροπο Σμίτ από την αρχή το επεξεργαζόμαστε καταβάλουμε πάρα πολύ μεγάλε προσπάθειε για να μην λησμονούμε αυτή την πτυχή. Δεύτερο πράγμα, στα πλαίσια του Erasmus Plus, είναι η υποστήριξη που θα δώσω αυτό το πρόγραμμα, θα ήθελα να συνεχιστεί. Σήμερα είναι 28%, αλλά όπω είπατε, χρειαζόμαστε αυτού του νέου, Αλλά τώρα έρχομαι στο τρίτο σημείο. Θα ήθελα, κατά τη διάρκεια του έτου, να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία που θα ήθελα να δημιουργήσει ευρωπαϊκό πλαίσιο μικροπιστώσεων είναι η εκμάθηση διαβίου, να αποκτά κανείς δεξιότητες όλη τη ζωή. Γνώση εμπειριών. Και θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτές, ούτω ώστε να βελτιώνονται οι προοπτικές, οι προσωπικές και οι επαγγελματικέ. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησα για τη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων. Θα δημιουργηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αυτή η ομάδα. Πρώτη συνεδρίαση προβλέπεται μέσα Μαρτίου θα τους δώσω 8 εβδομάδες, 8 εβδομάδες για να μου υποβάλουν μια έκθεση. Ξέρουμε ότι είναι ένα μοντέλο που υπάρχει, είναι ένα μοντέλο που άλλες χώρες εφαρμόζουν με μεγάλη επιτυχία. Εν συνεχεία το μήνα Μάιο στο Συμβούλιο θα υποβάλω μια πρόταση η οποία θα δημιουργήσει ευρωπαϊκό πλαίσιο για αυτές τις μικροδεξιότητες να λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή εμπειρίες και αυτά που μαθαίνει κάποιος. Θα πρέπει αυτή τη νέα μορφή να την αναλύσουμε. Και έρχομαι στο Digital Education Action Plan και επίσης τι θα, θέσεις θα έχει στα online courses, στην εκμάθηση στη διαδικτυακή. Να υπάρχουν μαθήματα στο διαδίκτυο, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν φυσικά. Και ερχόμαστε στο θέμα ποια είναι η αναγνώριση, ποια είναι τα πρότυπα, ποια είναι τα κίνητρα που δίνουμε. Και θα δούμε ότι στο Erasmus Plus εκεί θα επιμείνουμε, ώστε η, το διδακτικό ε, προσωπικό να έχει γνώσεις ψηφιακές, αν δεν αναγνωρίζει τα μαθήματα στο διαδίκτυο, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Συζητώντα τώρα με τους διδάσκοντες, βλέπουμε γιατί δεν έχουν κίνητρο να κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο, γιατί μετά δεν θα έχει ούτε αντίκτυπο ούτε στην καριέρα τους, ούτε στο μισθό τους να δίνουν μαθήματα στο διαδίκτυο. Σα διαβεβαιώνω ότι ένα θέμα το οποίο δεν λησμονώ. Αυτά τα τέσσερα πράγματα θα αναθίξω ότι έχει δρομολογηθεί και θα σας ενημερώνω δεόντως για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Λογόν Σφερόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σήμερα φτάσατε σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα λόγω του προπολογισμού. Αρκετά πράγματα, ερωτηματικά, αρκετά υπόθηκαν. Θέλαμε ο πολιτισμός και η παιδεία να μπει στο χαρτοφυλάκι, όσο σας δώσαμε μάχη. Δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι σήμερα ε, είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Να σας πω ότι δώσαμε τη μάχη σε επίπεδο συμβολικό μεταξύ άλλων και τώρα θα δοθεί η μάχη και σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να σας στηρίξουμε και να μας βοηθήσετε κι εσείς όμως. Να μας πείτε πώς συγκεκριμένα μπορούμε να κινηθούμε και να δράσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε, το, τη φιλόδοξη ατζέντα που μας παρουσιάσατε, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να έχουμε φιλοδοξίες ε, και να μην κινούμεθα και γρήγορα. Αλλά θα πρέπει να υλοποιούμε πράγματα εκτός των ονείρων. Και γι' αυτό έχουμε την απογοήτευση σήμερα. Αναφερθήκατε σε διάφορους στόχους να δημιουργηθεί και ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε το νέο Green Deal και της ψηφιακής Ευρώπης μεγάλα προγράμματα χωρίς να έχουμε έναν πλήρη χώρο να κινηθούμε. Και το βασικό θέμα είναι ο προπολογισμό στα χρήματα. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα, δεν υλοποιούνται τα προγράμματα. Αυτό που είναι δύσκολο στα πιο τεχνικά θέματα είναι αυτός ο κατεκερματισμός. Δηλαδή έχουμε το Erasmus Plus από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη έχουμε προγράμματα ερευνητικά Δημιουργούνται αρκετά ερωτηματικά πάνω σε αυτά. Μπορούμε να εξετάσουμε το δεχόμενο τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να μπορούν να ενδιαφερθούν από το ορίζον Ευρώπη. Υπάρχει μυστήριο επικρατή και υπάρχει μπλοκάρισμα όσον αφορά τα νέα προγράμματα. Διότι δεν υπάρχει περιεχόμενο και δεν υπάρχουν και αρκετά χρήματα. Και με τριπλασιασμό του Erasmus Plus που θα πετύχουμε ελπίζω, με δυσκολίε, αλλά γιατί όχι, να μην το πιστεύουμε, θα αρκούν τα χρήματα. Μπορούμε να έχουμε ε, κάποιες φιλοδοξίες στον φατοπροπολογισμό. Μαθητεία μετά. Επιμακρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε ευρωπαϊκό ε, χώρο μαθητείας. Δεν έχουμε ακόμα αναγνώριση των θεμάτων, των μαθημάτων. Ε, τι σημεία μπορείτε να στηρίξετε εσείς στο πρόγραμμά σας όσον αφορά αυτό το θέμα. Άλλο πολύ ενδιαφέρον που περιγράψατε για τη βασική εκπαίδευση. Η βασική διδασκαλία να προωθείτε; Πέρα από το να διαβάζει κανείς και να μετράει, είναι το θέμα της διδασκαλίας της ιστορίας. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Ξεκίνησε με τη δημιουργία του οίκου της ιστορίας, τη δημιουργία του παρατηρητηρίου Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Συζητείται αυτό το Σαββατοκύριακο το θέμα. Το θέμα του ε, σχολικού εγχειριδίου των βιβλίων των σχετικών στην Πολωνία. Είναι κάτι που αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Χωρί να επιβάλλουν στα κράτη-μέλη τι πρέπει να λένε, αλλά είναι το θέμα τη βασική διδασκαλία και το θέμα τη ιστορία για μένα είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το τομέα. Αύριο έχουμε σημαντική συνάντηση με του Υπουργού Παιδεία θα τους συναντήσετε πιστεύω, τι μήνυμα θα τους δώσετε. Θα συναντήσουμε ο καθένας με την Άννα, τους υπουργούς μας της παιδείας, ήδη τα όπως και με... μαζί με άλλους τους έγραψε επιστολές. Θα διαδώσουμε το μήνυμα, θα δώσουμε τη μάχη μας. Εσείς ε, τι θα κάνετε όσον αφορά την ευκαιρία αυτή που θα έχετε, τι μήνυμα θα δώσετε. Ευχαριστώ πολύ για τι ερωτήσει σα. Είμαι πολύ χαρούμενη που θέσατε το θέμα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη, διότι είναι ένα καλό παράδειγμα πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τον κύκλο εργασία. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση ΑΚ. Εδώ και μήνε λέω πόσο σημαντικό είναι η έρευνα και η καινοτομία να, από την αρχή να μπει στον κύκλο αυτό των πανεπιστημίων. Ήθελα να δείξουμε πόσο σημαντικό από την αρχή οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία με τις επιχειρήσεις, να δουν πώς προχωράνε τα προγράμματα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα, τα 5 εκατομμύρια ευρώ ε, δόθηκαν από την DG Γενική Διεύθυνση ΑΚ. Εδώ και δύο εβδομάδες πήρα την απόφαση τη διάσταση έρευνα και καινοτομία να τη βάλουν στις διάφορες συμμαχίες και γι' αυτό το λόγο το θέμα της μεταφοράς των πόρων χρειάζεται κάποια συνομιλίες με το Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, διότι υπενθυμίζω ότι στην Επιτροπή Ρέζη η μεταφορά των πόρων που στορίζονται Ευρώπη ε, σταμάτησε, μπλοκαρίστηκε. Ήδη μίλησαμε με τους συντονιστές, θα βρούμε μια λύση νόμιμη και ζήτησα από την ομάδα μου απλώς εμείς να δώσουμε το παράδειγμα, να δούμε πώς αυτές οι μεταφορές κονδυλίων μπορούν να γίνουν και ζήτησα να γίνουν μεταφορές κονδυλίων από τον ορίζοντα Ευρώπη προς τις συμμαχίες. Λοιπόν, τώρα μπορώ να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Το πρόγραμμα Horizon 2020, εκεί θα μεταφερθούν 2 εκατομμύρια ευρώ για κάθε μία συμμαχία, για να μπορέσουμε από την αρχή να συμπεριλάβουμε αυτή τη διάσταση της έρευνα και της ενοτομίας. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά καλά μαντάτα. Μετά είναι καθήκον μας η παρακολούθηση, διότι θέλουμε να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων, θα πρέπει να μας δώσουν ένα πλαίσιο πολύ πιο ευέλικτο και πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες. Νομίζω ότι θα χρειαστεί κάποια δεδομένη στιγμή να φροντίσουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να προχωρήσουμε αυτή η στατηγική μας για τη γνώση μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά τη μαθητεία και το πρόγραμμα των μαθημάτων, πιστεύω ότι θα πρέπει απλούστατα να επιληφθούμε περισσότερο επί του θέματος. Ποιος θα επεξεργαστεί αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων, εγώ είμαι πολύ ανοιχτή, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Από την πλευρά μου η ιδέα ήταν να έχουμε ευρωπαϊκό πλαίσιο μικρό μαθήσεων, διότι δεν είναι πάντα παραδοσιακά μαθήματα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι να αποκτήσουν εμπειρία και να αναγνωρίζεται η εμπειρία για να βρουν δουλειά. Το παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Ιστορίας δεν συνάντησε εκπροσώπους ακόμα, θα το κάνω αυτό, από την πλευρά μου το μήνα Μάρτιο θα είμαι στον οίκο της Ευρώπης ε, και θα το συζητήσουμε το θέμα. Ξέρετε ότι μέχρι τώρα έχουμε μόνο υλικό που διαδίδεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το υλικό Αντίθετα, γίνεται και διδασκαλία για την Ευρώπη. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και να δούμε μέχρι πού να προχωρήσουμε. Για ακόμη φορά, προσοχή όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και πόσο κόσμος θα το δεχτεί το θέμα. Ίσως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρούμε τη στιγμή να το κάνουμε αυτό. Θα μπορούσε να είναι θέμα ενός άτυπου γεύματο. Στα συμβούλια μπορούμε να το έχουμε αυτό για να δούμε ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Σήμερα δεν μπορώ να πω υπάρχει συνένεση μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είχα την ευκαιρία να το κουβεντιάσω με το κάθε κάτω μέλο αυτό το ζήτημα. Αύριο την Πέμπτη στο Συμβούλιο με τους υπουργού. πραγματικά πρέπει να πω το ότι είσαστε σε επαφή με τους υπουργού σας τους αντίστοιχους. Αυτό είναι πολύ θετικό, γίνεται αντιληπτό πολύ θετικά και έχει αντίκτυπο στη συνέχεια. Διότι με καλούν, μου λένε πώς αυτό το μήνυμα είναι σημαντικό και εκπλήσονται πολύ ευχάριστα, διότι ενώνει τη φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί τους. Αύριο θα συζητήσουμε το θέμα, διμερός, το θέμα του προπολογισμού, αλλά εν γέννη, όπως σας είπα, δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ για τον Υπουργό Παιδείας της Έρευνας και της Καινοτομίας. Οι Υπουργοί όλοι ε, μας στηρίζουν. Το πρόβλημα προέρχεται από εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις και ξέρουμε ότι είναι οι Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί Οικονομικών. Θέμα μας, βασικό θέμα, θα είναι το θέμα της κυκλοφορίας των εγκεφάλων. Ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την κρατική Προεδρία. Αυτό που μου αρέσει επίσης είναι το άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε μαζί του στη στιγμή του γεύματος. Να δούμε το, την Πράσινη Συμφωνία και τις αναγκαίες δεξιότητες και πώς η παιδεία μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία στόχο. Νέο θέμα, στην ανακοίνωση για το Green Deal υπάρχουν τρεις πτυχές οι οποίες υπογραμμίζονται πώ πώς μπορεί να συμβάλλει η παιδεία σε αυτά. Υπάρχει ποικιλομορφία στα διαφορα κάτι κράτη-μέλη, υπάρχουν διαφορέ. Και γι' αυτό χαιρετίζω τι πρώτε συζητήσει που θα έχω μαζί του και πραγματικά ανυπόμονα θέλω να ακούσω τι απόψει του, τι μπορούμε να κάνουμε, θέλουμε να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από κοινού, με κοινή προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άντερσεν. Είναι η τελευταία συντονίστρια και μετά έχουμε άλλους τρεις, αλλά έχουμε μόνο δέκα λεπτά. Οπότε κλείνει ο κατάλογος, ε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε με μετάφραση. Ωραία. Παρακαλώ. Ένα λεπτό ο καθένας ε, ε, στην ερώτησή του ε, η κυρία Άντρουσεν συντονίστρια έχει το λόγο και μετά οι υπόλοιποι για ένα λεπτό. Δυστυχώς σας περιορίζω, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων. Θα ήθελα ε, για τον εκπαιδευτικό χώρο του 2020 να μιλήσω. Η συνάδελφος Καμέβερ ε, ε είπε ότι συμφωνούμε ε, με το θέμα αυτό. Ε, έχουμε δει στην Γερμανία τα τελευταία χρόνια το ζήτημα του απολυτηρίου λυκείου και πώς ε, στην ουσία μας λείπουν τα εργατικά χέρια και έχουμε βάλει τα παιδιά μας σε μια απέλπιδα προσπάθεια για θέσεις εργασίας ενώ έχουμε εξαπατήσει και τους γονείς. Υπάρχουν παιδιά τα οποία τελικά ε, πληρώνουν ψυχιάτρους επειδή δεν πετύχανε στο πολιτήριο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε το image των ε, χειρονακτών και ε, πραγματικά σήμερα ενώ στο παρελθόν αυτά τα επαγγέλματα είχαν τόση φήμη, σήμερα κανείς ντρέπεται όταν έχει μια τέτοια δουλειά. καλό θα ήταν λοιπόν να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Τώρα, Θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας ε, και θα ήθελα να μάθω από σας συγκεκριμένα ως επίτροπος ε, θα κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε τα πανεπιστήμια της Ευρώπης ε, να διαδικτύουν να δικτυωθούν μεταξύ τους μάλλον. Ε, εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν ανταλλαγές, όμως όσον αφορά στα προγράμματα σπουδών, αυτό είναι θέμα της κάθε χώρας και έτσι πρέπει να μίλει. Καλό θα ήταν ε, λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά και γι' αυτό ζήτησα και το λόγο. Τέλος, να να σας μιλήσω για μία συνέντευξη που έγινε στις 29 Νοεμβρίου του 2019 στην Deutsche Welle και εκεί λέτε ότι ε, θα πρέπει να βάλουμε, δώσουμε έμφαση στις ικανότητες ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, για να μπορούν να συνταχθούν στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Όταν κάτι τέτοιο έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, καταλαβαίνετε ότι ε, το να έχετε στο παρελθόν ε, μειώσει τα χρήματα ε, για αυτά τα θέματα και να το γιορτάζετε ότι κάνατε εξοικονόμηση με βάση και τις πρακτικές της ΕΚΤ δεν συνάδει. Αυτό που δεν είπατε είναι ότι υπήρχε, υπήρχαν ε, πάρα πολλοί τόκοι που εισέπραξε το γερμανικό ε, κράτος τα τελευταία χρόνια, 368 ε, εκατομμύρια συγκεκριμένα, τα οποία δεν αναφέρθηκαν. Καλό θα ήταν λοιπόν να λέγονται τα πράγματα ότι ναι γίνεται εξοικονόμηση από την πλευρά της ΕΚΤ, όμως ε, στους πολίτες δεν λέμε ότι αυτοί πληρώσανε και βγήκαν αυτά τα κέρδη. Καλό θα ήταν λοιπόν στον ε, αγώνα της παραπληροφόρησης να σκεφτόμαστε και τέτοια πράγματα. Επειδή ε, θέλουμε όλοι οι συντονιστές να έχουν πάρει μια άμεση απάντηση. Θα απαντήσει τώρα η Επίτροπος και μετά οι υπόλοιπε ερωτήσεις θα πάνε όλες μαζί. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ε, δεν γίνεται διαφορετικά. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ε, καταρχάς, για το θέμα της επαγγελματική εκπαίδευσης, εν μέρει έχω ήδη απαντήσει, απλώς να προσθέσω εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, Εμεί συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Τιερή Μπρετών, ο οποίος ε, θα ξεκινήσει μια νέα βιομηχανική πολιτική και όλα τα industrial skills, τα βιομηχανι... τις βιομηχανικές ε, δεξιότητες που ε, θα, προωθήσει, θα τις προωθήσω και εγώ. Υπάρχουν και τα blueprint skills που είναι ένας άλλος τομέας που μας ενδιαφέρει. Δεν τα χάνουμε από το, από το βλέμμα μας αυτά. Επίσης, είναι πολύ σημαντικές οι ψηφιακές δεξιότητες, γιατί όλες αυτές οι μηχανές που βρίσκονται στους παραδοσιακούς ε, βιομηχανικούς τομείς ε, σήμερα χρειάζονται ανθρώπινο έλεγχο και δεν πρέπει κανείς να χάσει τη σύνδεση, αλλά πρέπει να είμαστε και ανοιχτοί ε, στην ψηφιακή εποχή, ακόμα και στους πιο παραδοσιακούς τομείς που γνωρίζουμε, συγκεκριμένα με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εντάξει, οι μεγάλοι έχουν την ανάγκη και κάνουν πράγματα, αυτές βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Τώρα, για την παραπληροφόρηση, μέσα στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Αυτά ζήτησαν να συμμετάσχουν, αυτά ε, στην ουσία μπήκαν μπροστά και μας είπαν στα τρία χρόνια αυτά να τα εμπόδια να τι μπορούμε να κάνουμε. για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι να μην αναπαράγουμε τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Δεν χρειαζόμαστε τώρα και πάλι projects ε, που τα τρέχουν 3, 5, 7 χώρες. Ε, πρέπει να σκεφτούμε την ηλεκτρονική κάρτα του φοιτητή, πώς να υπάρχει πρόσβαση στις εταιρείες, ε, πώς μπορεί να δίνεται η δυνατότητα Έβρεση εργασίας ήδη από την εποχή του πανεπιστημίου. Όμως τα πανεπιστήμια πρέπει να μας το πούνε πώς θα το κάνουμε, πώς θέλουν να είναι το μέλλον και αυτό δυστυχώς δεν μας ε, καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουμε θέματα περίπλοκα, ειδικά αν τώρα ε, υπάρχουν τέτοια θέματα που ανακύπτουν όπως ας πούμε το καθεστώς των πανεπιστημίων κτλ. Έχουμε λοιπόν όλη αυτή την ελευθερία που δίνουμε στα πανεπιστήμια γιατί είναι ανεξάρτητα και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Τέλος, για το media literacy. Ε, είναι ένα θέμα που το θέλω ε, πολύ να το προωθήσω γιατί αυτός ο αγώνας κατά της παραπληροφόρησης περνά από την υπευθυνότητα των πλατφορμών αλλά πάνω απ' όλα είναι η εκπαίδευση, η κριτική σκέψη που θα επιτρέψει στα παιδιά μας να κάνουν επιλογές. Όταν ξεκίνησα τον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης ήμουν ξεκάθαρα. Υπάρχουν δύο κόκκινες γραμμές. Ε, η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία. Αυτές δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Πρέπει να δώσουμε όμως τα εργαλεία στους νέους για να μπορέσουν ελεύθερα να κάνουν την επιλογή τους. Γι' αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένη που αυτή τη φορά η μάχη κατά της παραπληροφόρηση στους νέους έχει πέσει στα δικά μου χέρια και μέσα από τα πλαίσια του Digital Education Action Plan θα λάβω πρωτοβουλία σας. Θυμίζω ότι υπάρχει και η πρωτοβουλία Safer Internet for EU. Ε, για... Ξεκίνησε το 2019 και έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ε, Ευρωπαίους πολίτες που συμμετέχουν οι νέοι για μένα είναι σημαντικό να μην ακούν μόνο τι πρέπει να κάνουν, αλλά να έχουν τα εργαλεία για να επιλέγουν μόνοι τους. Και ειλικρινά θα είμαι περήφανη αν οι πρωτοβουλίες που ξεκινήσαν πέρυσι με το European Media Literacy Week συνεχίσουν, γιατί υπήρξε η πρώτη έκδοση είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ και από την πλευρά μου θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον Επίτροπο Μπρετών για να μπορέσει να συνεχίσει αυτή η πρωτοβουλία και για να μπορούμε παντού στο χάρτη της Ευρώπης να βλέπουμε νέους που μπορούν να ε, δραστηριοποιούνται ενεργά σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη σειρά ομιλητών. Σας ζητώ να είστε πολύ σύντομοι. Αντέμοφ, Μπλάνκο και Σεκουρέλ. Αυτοί είναι οι επόμενοι ομιλητές. Ένα λεπτό, θα είμαι πολύ αυστηρή. <clears throat> Κύριε Επιτροπέ, στην αρχή της εισαγωγής σας είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε φιλόδοξου, έχει φιλόδοξους στόχους σήμερα και για να επιτευχθούν χρειάζονται πόροι και οικονομικοί αλλά και ανθρώπινοι πόροι. Εκεί λοιπόν έρχεται να παίξει το ρόλο του το εκπαιδευτικό σύστημα. Το απόγευμα θα συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, το AI, τεχνητή νοημοσύνη. Ε, έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις. Είναι αυτονόητο ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ε, θα επωφελήσει το εκπαιδευτικό σύστημα, όμως υπάρχουν ταυτόχρονα κίνδυνοι που παραμονεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που θα χάσουν, ε, για παράδειγμα, τη δουλειά τους. Οι δάσκαλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να ανοίξουν τον δρόμο για τα νέα επαγγέλματα του μέλλοντος. Υπάρχει κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει και κενό μεταξύ των μικρότερων και μεγαλύτερων περιοχών. Ευχαριστώ κύρια Επίτροπε. Θα ήθελα να σχολιάσω ένα από τα θέματα που αναφέρατε. Η πρότασή μας για την νέα διαχείριση του προγράμματος δεν σημαίνει ότι θέλουμε να χαλάσουμε τη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Απλώς θέλουμε μια φυσιολογική σχέση. Να δώσουμε πνοή σε μια φυσιολογική σχέση. Έτσι κατάλαβα από αυτά που είπατε εσείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι κάποια ευρωπαϊκή κυβέρνηση, είναι ένα εκτελεστικό όργανο ε, που ε, εκτελεί τα νομοθετήματα δύο νομοθετών, δύο θεσμών. Όμως ε, θα πρέπει να παίξετε κι εσείς αυτό το ρόλο, σύμφωνα με το, αυτή τη δομή. Ευχαριστώ πολύ ως προς την ανακοίνωση που κάνατε για την εγγύηση για τους νέους, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Θέλω να τονίσω ότι έχει ενσωματωθεί στη Συμφωνία του Γκέτεμπορκ, την εγγύηση για την παιδική ηλικία. Ένας από τους πυλώνες της εκπαίδευσης, ε, άλλος πυλώνας ήταν η διατροφή, ε, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σε καταστάσεις υγειονομικής προστασίας ε, και στέγαση, εκπαίδευση, οικογένεια κτλ. Θέλω να τονίσω το εξής. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε μόνο ψηφιακές διεξιότητες. Είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση και φιλοσοφική προσέγγιση. Το να καταλάβει κανείς τι ακριβώς σημαίνει ε, αυτή η πολιτισμική αλλαγή που θα βιώσουν οι κοινωνίες μας ε, στο μέλλον με την ε, επικράτηση της ψηφιοποίηση. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτές τις δύο προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολας Νένας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε και Επίτροπος Πολιτισμού και σας ευχαριστούμε που ξαναβάλατε την λέξη αυτή στον τίτλο. 80% των αιτήσεων για το πρόγραμμα το πολιτιστικό δημιουργική Ευρώπη δεν μπορούν να τύχουν ικανοποίησεις γιατί απουσιάζει χρηματοδότηση. Και εκεί συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσει που εκκρεμούν από προηγούμενα, γιατί οι διαχειριστές λένε σας παρακαλώ μην υποβάλλετε άλλη αίτηση για χ πρόγραμμα γιατί δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί. 6,9% λιγότερο είναι η πρόταση. Πτώση. Ποια είναι η άποψή σα, τι, πρέπει να γίνει για να αυξήσουν τα κράτη-μέλη τον προπολογισμό αντί να τον περικόπτουν. Είναι κοινό μα μέλημα και επιδίωξη Επιτροπή και Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Η κυρία Σικουρέλ, παρακαλώ. Καλημέρα και πάλι. Είναι η πρώτη συνεδρίαση εργασία για μένα, παρουσία δική σα και είμαι και εγώ συγκινημένη που είστε εσεί εδώ. Θέλω να εκφράσω την οργή μας και εσείς ημερίζεστε την δωρική μας και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Το Εράσμος δεν μπορεί να είναι θέμα προεκλογικής εκστρατεία από τη μία και να το έχουμε λάβαρος προεκλογικές εκστρατείε και μετά να το ρίχνουμε στα τάρταρα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε το Εράσμος Plus και οι φιλοδοξίες μας να τεθούν στο περιθώριο. Εμείς θέλαμε να διευρύνουμε το Εράσμος, να αγγίξει και άλλες πληθυσμιακές ομάδες ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο εν ώψη των καταιγιστικών εξελίξεων της παγκοσμιοποίησης. Ε, όσοι θέλουν να το περικόψουν δείχνουν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα για το δημοκρατικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε όλοι. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Ποια είναι η γνώμη σας για ένα τεράστιο σχέδιο δράσης για τα fake news. Είναι και δικιά σας προτεραιότητα. Θα ήταν ευπρόσδεκτο ένα τέτοιο σχέδιο. Και επίσης, Ποια είναι η γνώμη σας να σταματήσουμε πλέον να μιλάμε για κόστος της εκπαίδευσης, αλλά για επένδυση στην εκπαίδευση. Ναι, έχουμε ξεπεράσει τα πέντε λεπτά που μας έδωσαν οι διερμηνείς. Ε, επειδή λοιπόν θα φύγουν οι διερμηνείς μας, πρέπει να γυρίσουμε στα αγγλικά για την απάντηση. Ε, μάλλον ξεκινήστε και όταν ε, πούν για οι διερμηνείς, κλείνετε Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ τους διερμηνείς. Ε, ε, δεν χρειάζεται να το πω ε, πολλές φορές. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό δεν είναι απλώς επενδύσεις σε χρήματα, είναι επένδυση στο μέλλον μας. Είναι κομμάτι της δημόσιας δήλωσης κάποιων άλλων, όμως τώρα αυτό που βλέπετε εσείς να δείτε είναι οι πράξεις και τα γεγονότα. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της ε, ψηφιακής τεχνολογίας. Εκεί πρέπει να είμαστε ε, υπέρ μιας ολιστικής ε, προσέγγισης, όχι μόνο στις δεξιότητες αλλά και στην υποδομή για το Digital Education Action Plan. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα ε, σχολεία να έχουν υψηλής ταχύτητας ε, ίντερνετ, ε, γιατί στο Erasmus Plus μιλάμε για τεράστια εγχειρήματα και τα σχολεία δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες. Πρέπει να φροντίσουμε μέσα στα πλαίσια του Green Deal οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει, τα 3 δις ευρώ να δοθούν και για την, να εξοπλιστούν τα σχολεία μας με την υποδομή που χρειάζεται. Πόσο μάλλον που έχουμε τη δυνατότητα ε, γιατί ήμουν εδώ όταν ε, είχε τεθεί αυτό το θέμα. Μιλήσαμε για την ψηφιακή υποδομή, μιλήσαμε ε, για την ανάγκη να υπάρχουν ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους διδάσκοντες για να μπορέσουν να εμπνεύσουν τους νέους. Η τεχνητή νοημοσύνη, θα είμαι ξεκάθαρος, ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον οποιονδήποτε. Τα ανθρώπινα όντα πρέπει να είναι εκεί και να ε, έχουν τον έλεγχο. Σας ε, αφυπνίζω λοιπόν ενώπιον αυτού του κινδύνου. Στη Λευκή Βίβλο το λέει ξεκάθαρα η ευρωπαϊκή προσέγγιση δεν είναι ούτε αυτή των ΗΠΑ ούτε της Κίνας γιατί στη δική μας περίπτωση εμείς θέτουμε την αξία στις ηθικές μας αξίες. Ναι, υπάρχει κίνδυνος, κίνδυνος ε, κάποιων ε, προκαταλήψεων, ε, ακόμα και διακρίσεων, όμως εμείς δεν θέλουμε την αναγνώριση προσώπου. Ξέρετε ότι υπάρχει στην Κίνα και σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα πάνε πολύ πολύ μακριά. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί καταρχάς να απαντά σε ξεκάθαρες απαιτήσεις στην ασφάλεια, στις αρχές, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και μετά να θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει η τεχνητή νομοσύνη. Θα μπορούσε ας πούμε να είναι πιο χρήσιμη για να είναι πιο προσωποποιημένη η σχολική σταδιοδρομία. Ε, ας πούμε σε μια τάξη με 30 παιδιά, έχουμε κάποιους που πάνε πιο γρήγορα, κάποιοι άλλοι που πρέπει να προσαρμόσουμε ε, την εκπαίδευση στις δικές τους ανάγκες. Ε, επίσης υπάρχει και αυτό το χάσμα μεταξύ των αστικών και μη περιοχών. Δεν πρέπει να τα χάνουμε αυτά από το βλέμμα μας. Τέλος, για το Creative Europe δεν σταματώ να το λέω όπου και αν πηγαίνω, σε όποια χώρα. Θα πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει μικρή συμμετοχή γιατί απλώς δεν υπάρχει εθνικός μηχανισμός συγχρηματοδότησης. Όσοι δεν έχουν θα το, θα το αποκτήσουν. Επίσης υπάρχει και η συμμετοχή τρίτων χωρών. Υπάρχουν νέοι μηχανισμοί για το πρόγραμμα Media. Έχουμε πει ότι θα ε, σεβαστούμε τις, τους νέους ε, μηχανισμούς ε, της Οδηγίασε για τα οπτικοακουστικά μέσα. Ε, αυτά δεν γίνονται αυτόματα. Επίσης, ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέχουμε όταν διευρύνουμε αυτή την πρόσβαση το είπα τον Σεπτέμβρη και δεν έχω αλλάξει. Δεν θα βασιστώ μόνο στο Creative Europe, αλλά και στο κίκ στις ε, ε, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Μιλάμε για 3 δις ευρώ. Κάντε τη σύγκριση με το κομμάτι του πολιτισμού του Creative Europe. Στο δεύτερο πυλώνα του Horizon Europe θα έχουμε ε, ένα κομμάτι που θα είναι ακριβώς για το δημιουργικές αυτές βιομηχανίες. Αυτά τα projects που δεν πήραν χρηματοδότηση από το Creative Europe επειδή υπήρχαν άλλες απαιτήσει, πώς θα έχουν πιο άμεση πρόσβαση. Τέλος, για τα fake news, το ευρύτερο ε, σχέδιο ε, το επεξεργαζόμαστε. Η Επίτροπο Γιούροβα είναι υπεύθυνη. Εγώ από την πλευρά μου είμαι υπεύθυνη για την πάταξη τη παραπληροφόρηση μέσω τη εκπαίδευση, μέσω τη νεολαία, ε, το critical thinking, media literacy. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς, το μεγαλύτερο ίσως ε, που βρίσκεται στα δικά μου χέρια. Και επίσης εμείς είμαστε για πρώτη φορά στη θέση να έχουμε τα μέσα. Σε ένα διατομεϊκό κομμάτι, συγγνώμη, θα πρέπει να συνεχίσετε στα αγγλικά, γιατί οι διερμηνείς ε, θα φύγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διερμηνείς που έμειναν 11 λεπτά παραπάνω. Σας ευχαριστούμε και οι διερμηνείς σας ευχαριστούν. And we continue for the rest of the answer in English now. Thank you.